Δεν μπορούμε να φύγουμε από εδώ από το 2Q2. So I'm very glad that... Πάλι εδώ. Και πάντως κάποιοι από εσά μείνανε. Και είναι εδώ παρόντες. Άρα να ξεκινήσουμε το δεύτερο τμήμα της συνεδριάσεως, την απογευματινή συνεδρίαση της Επιτροπής μας. Το πρώτο σημείο σήμερα σε διάταξη τώρα, ή το 13ο τέλο πάντων από την αρχή, είναι οι ευκαιρίε τη πράσινη ανάπτυξη για τι μικρομεσαίε επιχειρήσει. Είχαμε και πριν την ευκαιρία να συζητήσουμε για τι μικρομεσαίε επιχειρήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με την ενέργεια και τι ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια. Και τώρα έχουμε την να συζητήσουμε για τι ευκαιρίε πράσινη ανάπτυξη. Με εισηγητή τον Φίλιπ Ντεμπάκερ. Κατόπιν της ανακοίνωσης της Επιτροπής για το πράσινο πρόγραμμα δράσης, το οποίο δημιούργησε ένα πλαίσιο για να δούμε τι ευκαιρίε μπορεί να υπάρξουν για να εκμεταλλευτούν να ΜΜΕ. Για το πώ θα ενεργήσουν, πώ θα δράσουν, πώ θα κινηθούν οι ΜΜΕ και μην ξεχνούμε ποτέ για το πόσο βοηθούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσει για την επαναβιομηχάνηση τη Ευρώπης. Η επαναβιομηχάνηση της Ευρώπης, πολύ σημαντικό. μια τρομομηχανή για την ανάπτυξη και την πρόοδο της Ευρώπης. Για μια οικονομία βιώσιμη και ανταγωνιστική. Όλα αυτά τώρα να συζητήσουμε και επίσης θα πρέπει να προγραμματιστούμε σε σχέση με την μετάβαση στην πράσινη ανάπτυξη και πώς θα ωφεληθούν οι ΜΜΕ από την ε, δοσματική χρήση των ανηδιακών πόρων. Κύριε θέλω θα μας προσθέσετε τις απόψεις σας. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ για την ευκαιρία αυτή για να επεκταθώ λίγο όσον αφορά τι ιδέε, τι προτάσει μου, αλλά θα έχω και την ευκαιρία να ακούσω και του αδέλφου για να μάθω και τι δικέ του απόψει για το πώ θα εξελιχθεί αυτή η έκθεση. Ο, η ιδέα αυτή για την πράσινη ανάπτυξη είναι να εκμεταλλευτούμε τι επιχειρησιακές, επιχειρηματικές ιδέε που υπάρχουν που παρουσιάζονται με αφορμή τη μετάβαση σε μια πιο βιώσιμη οικονομία, έχουμε όλο ένα και μεγαλύτερο πληθυσμό, έχουμε όλο ένα και περισσότερη ανάγκη για πρώτες ύλε. οπότε και θα πρέπει να βοηθήσουμε να προσαρμοζούν σε αλλαγέ οι επιχειρήσει και στον τρόπο λειτουργία του. Ακόμα καταναλώνουμε πολλά και τότε θα χρειαστούμε, αν συνεχίσουμε αυτό, το επόμενο 20 ετία έχουμε 40% περισσότερη ενέργεια που ξέρουμε ότι αυτό δεν είναι α, κάτι το α, βιώσιμο. Επομένως, μακροπρόθεσμα δεν είναι δυνατόν να συνεχίσουμε έτσι. Και μπορούν οι συνάδελφοι να δείξουν μια την για το τι λέω όσον αφορά για μια οικονομία χαμηλών εκπομπών. Αλλά επίσης έχουμε τώρα και τις κατάλληλες ε, συνθήκες για την καινοτομία, ώστε να μπορούν οι εταιρείε να μεταλλευτούν ε, τις ευκαιρίες από αυτήν την αλλαγή. Εξορισμού είμαι λογικός είμαι φιλελεύθερος και κυρίως αισιόδοξο. Οπότε να δούμε τώρα τι ευκαιρίες παρουσιάζονται, ας πούμε, τι γίνεται στην παγκοσμία αγορά, για τα περιβαλλοντικά αγαθά. Μιλάμε για ε, ένα τρεις και αυτό μπορεί να τριπλασιαστεί μέχρι το 2020. Μιλάμε για ένα ποσό το οποίο μπορεί να φτάσει ε, να τριπλασιαστεί, ε, να τριπλασιαστεί σε σχέση με το κεφάλαιο επενδύσεων της πρότασης Juncker. Έχουμε επομένω το ανάπτυξη τη πράσινη οικονομία, οπότε και αυτό επίση συμβάλλει στην ανάπτυξη αυτή και θα πρέπει να δούμε πώ θα εξωθήσουν προ αυτή τη κατεύθυνση του Ευρωπαίου ηγέτε. Και έχουμε κάποιε εταιρείε που επενδύουν σε αυτή την οικονομία, είναι δραστηριε και αυτέ επίση αποτελούν δυνατότητε για το μέλλον και να είναι η βάση τη βιομηχανία την επόμενη δεκαετία. Επομένως ό,τι κάνουμε θα αφορά τους ε, φευρέτες, τους ερευνητές, αλλά θα πρέπει να τους δώσουμε το κατάλληλο πλαίσιο να εκκίνηθουν. Αυτή είναι η βάση της ε, έκθεσης, το τι είδος πλαίσιο θα πρέπει να δημιουργήσουμε για αυτούς. Όλο ένα και πιο βασικό είναι αυτό στα γραφτά των οικονομολόγων, αυτή η πράσινη ανάπτυξη. Να βοηθήσουμε την ανάπτυξη την ε, εκμετάλλευση των πόρων, μείωση της μόλυνσης σε αέρα, γη και θάλασσα και όλα αυτά θα πρέπει να συνδυαστούν με την αναζήτηση της ανάπτυξης και την ανάγκη να υπάρχει μια ανάπτυξη που να είναι αηφόρος. Έχουμε πολλές απώλειες όμως σε αυτή την πορεία που κάνουμε είναι το τι έχουμε δημιουργήσει, το τι έχουμε μάλλον διαθέσει για την ε, παραγωγή. Και συνήθως αυτό το οποίο κάνουμε είναι να επεμβαίνουμε εκ των υστέρων. Μπορεί όμως ότι, έχει, ότι είναι απώλεια ενός εργοστασίου να χρησιμοποιηθεί σε ένα άλλο. Άρα να δούμε πώς θα χρησιμοποιήσουμε όλο ένα και λιγότερες πρώτες ύλες ή πόρους. Πιο οικονομική η πορου πιο οικονομικη παραγωγής με σύγχρονες τεχνολογίες και έτσι θα μειώσουμε την εξάρτησή μας από εξωτερικούς παράγοντες και αυτό ισχύει για όλα τα εμπορεύματα, τις πρώτες ύλες, τους ενεργικούς πόρους. Με αυτή την αλλαγή στις παραγωγές θα έχουμε να φέρουμε το, θα μειώσουμε το, το κόστος της παραγωγής και την εξάρτηση με. Έχουν πολλές χώρες που έχουν ακολουθήσει μια τέτοια στρατηγική και αυτή είναι τα παραδείγματα προς μίμηση. Έχουμε επίσης πολλούς άλλους τρόπους που μπορούν οι εταιρείε να συμβάλλουν στο πώς θα γίνει πράσινη η οικονομία μας. Να γνωρίζουμε τα σχετικά με την ενέργεια. Αλλά θέλω να καταλήξω την παρουσίαση όσον αφορά της ΜΜΕ, το δεύτερο τμήμα δηλαδή της έκθεσης. Τα ξέρετε να μην τα επαναλάβω, κάναμε και χθε ε, την ακρόαση και ήταν ξεκάθαρο το τι ρόλο μπορεί να θερματίσουν οι ΜΜΕ. Και επίσης ε, ακούσαμε από πρώτο χέρι τι γίνεται που αφορά τις ε, ε, ΜΜΕ. Τελικά το θέμα είναι βέβαια το να έχουμε ένα καλό περιβάλλον, περιβάλλον επιχειρηματικότητας, για αυτές τις καινούργιες μειωσερχόμενες στην αγορά έψιλο, να έχουν τις κατάλληλες ευκαιρίες. Άρα ευκαιρίες, λιγότερη γραφειοκρατία, κατάλληλη νομοθεσία και να αρθούν οι φραγμοί για αυτές τις μικρές εταιρείες. Προσβασιμότητα επίσης στο δανεισμό, στο κεφάλαιο που το βασικό πρόβλημα, εκτός από την γραφειοκρατία. Επίσης θα πρέπει να έχουμε κάποιο είδους ε, προγράμματα επιχειρηματικά και έτσι να ρίξουμε στον τομέα αυτό χρήμα. Επιχειρηματικό πνεύμα το οποίο πρέπει να τονωθεί. Να ολοκληρώνει την ιστορική αγορά μέσω καταλήλων ε, συμβάσεων και να δούμε πώς αυτές οι εταιρείε μπορούν να λειτουργούν πιο εύκολα, πώς μπορούν να προχωρήσουν σε αυτή τη νέα φάση της οικονομίας και να δούμε το πώς θα εκμεταλλευτούν οι ΜΜΕ τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται από την πράσινη ανάπτυξη. Νομίζω ότι με αυτή την έκθεση και την πλήθεια των συναδέλφων θα στείλουμε το μήνυμα σε Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά το τι ενδιαφέρει εμάς ως Ήτρα. Ευχαριστούμε κύριε Σιγητά. Τώρα είσαι σχεδόν Σιγητά. Εκ του ΕΛΚΟ, κύριο Ρούμπιχ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και τον εισηγητή. Φίλιπ Τιμπάκερ. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ θετικό το γεγονός ότι θέτουμε στο επίκεντρο την ανάπτυξη Πράσινη ανάπτυξη για μένα τι σημαίνει ότι θα πρέπει τα φανάρια να ανάψουν στο πράσινο. Θα πρέπει να είναι λοιπόν δυνατόν να μπορέσουμε να τοποθετηθούμε στην ε, αιχμή του δόρατο σε ό,τι αφορά την τεχνολογία. Γι' αυτό λοιπόν η πράσινη ανάπτυξη είναι η ανάπτυξη η οποία θα δημιουργήσει θέσει εργασία, κυρίω για του νέου. Και έτσι όχι μόνο στο ιστορικό αλλά και στο εξωτερικό της ε, Ευρώπης θα έχουμε ευκαιρίες. Θεωρώ ότι η πολιτική ανάπτυξη έχει πολλές δυνατότητες για μας που θα ανοίξουν στην Μεγάλη Αφρικανική Ήπειρο όπου πολλές υποδομές ακόμα είναι απαραίτητες σε ό,τι αφορά θέματα υγιεινής, άδευσης, ίδρευσης, αποχέτευσης, βιομηχανίας και το καθεξής. Και σε ό,τι αφορά τις ε, συγκρούσεις που συζητιώνται. Θεωρώ λοιπόν ότι φέρουμε ευθύνε όχι μόνο για την Ευρώπη αλλά για τις παγκόσμιες εξελίξεις και γι' αυτό λοιπόν είναι τόσο σημαντικό το θέμα της έκθεσης. Πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα ελκυστικό επενδυτικό κλίμα για την επαναβιομηχανοποίηση της Ευρώπης. Ο πρώην Επίτροπος Ταγιάννη δήλωσε ότι υπάρχει ο στόχος του 20% μέχρι το 2020 σε θέματα ενεργειακών και κλιματικών στόχων. Φαίνεται ότι θα πετύχουμε τους στόχους μας, αλλά μόνο στην επαναβιομηχανοποίηση, στη δημιουργία θέσεων εργασίας φαίνεται ότι δεν τα πηγαίνουμε καλά. Μείον 1,8% Μειώσαμε δηλαδή το 15,5% στην Ευρώπη και τα 1,8%. Και υπάρχουν χώρες που δεν ε, είχαν σωστή βιομηχανική πολιτική όπως η Ελλάδα για παράδειγμα με 11% ή η Γαλλία με 12-13%. Εδώ πέρα λοιπόν υπάρχει κατεπηγόντως ανάγκη να κάνουμε κάτι. Θα πρέπει στην Ευρώπη να μπορούμε να παράγουμε την ενεργειά μας ανά έτος 5 δισεκατομμύρια δαπανάμε για να αγοράζουμε ενέργεια. Αναρωτιέμαι λοιπόν γιατί δεν μπορούμε πιο πολύ ενέργεια με ευνοϊκότερους όρους και ευνοϊκότερες συνθήκες να την παράγουμε στην Ευρώπη. 200 δισεκατομμύρια ευρώ αγοράζουμε κάθε χρόνο σε πρώτες ύλες. 7 δισεκατομμύρια δηλαδή μιλάμε. Ξεπερνάει λοιπόν το πρόγραμμα του Ιούνκερ κατά πολύ το ποσό αυτό. Θα πρέπει όμως λοιπόν να περάσουν όλα αυτά, να εφαρμοστούν σε πολιτική όχι μόνο ε, η προστασία της φύσης, είναι θετικά τα μέτρα Natura 2000 των φυσικών βιότοπων, αλλά θα πρέπει να δημιουργήσουμε κάτι ανάλογο. Θα πρέπει να υπάρχουν προστατευόμενες βιομηχανικές περιοχές. Περιοχές όπου θα μπορούμε να εργαζόμαστε. Θεωρώ ότι η μακροπρόθεσμα, η στρατηγική και ο στρατηγικός σχεδιασμός σε ό,τι αφορά την χορταξία θα πρέπει να προβλέπει και χώρους όπου θα δημιουργούνται νέες θέσεις απασχόλησης και ο πρόεδρος ε, με κοιτάει ανήσυχο. Αλλά ο κύριος Τατζάνη νομίζω δεν έχει έρθει ακόμα. Και για να αποφύγω τις ε, παύσεις, σκεφτήκα να καλύψω την ε, παύση. Ναι, είναι εδώ όλοι οι σκιώδες όμως. Καλά λοιπόν, σταματάω, πρόεδρε. Λέει ο κύριος Ρουμπίχη. τελείωσα. Σας ευχαριστώ, λέει ο πρόεδρος, σας ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Κόφοντς, από τους Σοσιαλιστές και Δημοκράτες. Ευχαριστώ, πρόεδρε, ευχαριστώ και τον εισηγητή Είναι οπωσδήποτε μια πολύ καλή ευκαιρία αυτή για να συζητήσουμε την έκθεση και να καταλήξουμε σε μια αποτελεσματική ε, οικονομία απαλλαγμένη από άνθρακα με νέες συνθήκες, προϋποθέσεις για θέσεις εργασίες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις αλλά και επαναβιομηχάνηση της οικονομίας της Ευρώπης. Νομίζω ότι είναι από τα πιο σοβαρά πράγματα που μπορούμε να κάνουμε για να υπάρξει μια πράσινη μετάβαση στην Ευρώπη. Αυτή θα ήταν η επί της ουσίας ευκαιρία. Συμφωνώ μαζί σας και με τον εισηγητή και απλώς να προσθέσω κάποια πράγματα, διότι αν δούμε την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, επικεντρώνεται ιδιαίτερα στις μικρομεσαίες. Όμως πρέπει να μας απασχολήσουν και οι μικροεπιχειρήσεις, αλλά και οι νεοσύστατες. Πρέπει να δημιουργήσουμε ε, και να καλλιεργήσουμε ένα πνεύμα επιχειρηματικότητα στην Ευρώπη. Νομίζω είναι πολλές οι επιλογές να δώσουμε κίνητρα. Λόγω χάρη όταν κάποιο ξεκινά μια νεοσύστατη εταιρεία, η πρόσβασή του στην αγορά πρέπει να διευκολύνεται και αυτά θα πρέπει να γίνουν κανόνες στην Ευρώπη. Ε, Γιατί την ε, διατομιακή συνεργασία. Εταιρείε από διαφορετικούς κλάδους θα πρέπει να μπορούν να έχουν κοινά συστήματα διαχείρισης αποβλήτων λόγου χάρη ή πρώτων υλών. Στη χώρα μας, Τη Δανία, έχουμε πολλά καλά παραδείγματα για το πώς μπορεί να λειτουργήσει ένας τέτοιο συντονισμός. Και τρίτον, το χάσμα της γνώσης, της τεχνογνωσίας. Πρέπει να καλυφθεί το κενό αυτό, διότι πολλές εταιρείε δεν έχουν αρκετούς πόρους Είναι πολύ σημαντικό πώς οι πόροι αυτοί θα επαναχρησιμοποιούνται ή θα αξιοποιούνται. Πρέπει να μας απασχολήσει το θέμα και των συντονιστών, διευκολυντών, όπως τους πούμε, τους ε, ε, επιτραμμένους επί του συντονισμού σε τοπικό επίπεδο είναι πολύ σημαντικό και αυτό και από τα τελευταία ταμεία, την ΕΤΕ, το Horizon 2020 πρέπει να αναζητήσουμε πηγές και αναβάθμιση στο κατασκευαστικό τομέα με τα τούβλα, τα παράθυρα, τα κουφώματα, τις στέγες, όλα αυτά πρέπει να αξιοποιηθούν. Πρόεδρε, σας βλέπω, ξέρω ότι εξαντλεί το χρόνος μου, αλλά είναι πολλές ιδέες που έχουμε, έχουμε πολλά να πούμε και να σκεφτούμε λίγο και τις μεγαλύτερες εταιρείε. Αυτές που έχουν ενεργειακή, μάλλον καλή διαχείριση των πόρων τους. Οι εταιρείε αυτές είναι αυτές που είναι ψηλά στην αλυσίδα της ε, αξίας και με τις εξαγωγές τους φέρνουν εισόδημα στη χώρα. Αυτή λοιπόν την αλυσίδα ποιότητας να την προωθήσουμε, όπως είπατε και εσείς στις αγωγικές σας παρατηρήσεις. Ανυπομονώ λοιπόν να συνεργαστούμε στενά με τον εισηγητή από τους Σοσιαλιστές και Δημοκράτες. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Κόφωτ. Κύριε Ζούλο. Εδώ είμαι. Ευχαριστώ. Να ξεκινήσω τα δεδομένα που παρουσιάζονται από το πράγμα δράση για τι μικρομεσαίε επιχειρήσει. Βλέπουμε εδώ ότι 93% των μικρομεσαίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήδη έχουν πρωτοβουλίε για αποτελεσματικότερη χρήση των πόρων ή τουλάχιστον το επιδιώκουν. Το 42% έχει πραγματικά αποτελέσματα. Αποτελέσματα στην πράξη από αυτές τις πρωτοβουλίες, από αυτές τις ε, απόπειρες. Αυτό σημαίνει ότι το πρόβλημα είναι το εξής. Τα μέσα που χρησιμοποιούνται ε, θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν, όμως δεν είναι καθόλου αποτελεσματικές ή νομοθετικές πρωτοβουλίες. Θα πρέπει λοιπόν να στοχεύουμε στο να γίνουν πιο εύχριστες οι πρωτοβουλίες μας προτάσεις για να βελτιωθεί η πρόσβαση στα κονδύλια, συμμετοχή των αρχών τοπικής αυτοδίκησης, που θα μπορούσαν να ευνοήσουν την δικτύωση, την... τον συντονισμό και την πρόσβαση των μικρομεσαίων σε αυτές τις πηγές χρηματοδότησης. Και κάτι που για μένα είναι ακόμη πιο σημαντικό είναι να εφαρμοστεί μια προσπάθεια παρακολούθησης των αποτελεσμάτων διαρκής, διότι κατά αυτόν τον τρόπο θα μπορούσαμε να είμαστε και ε, ταχείς στην διόρθωση των προβλημάτων και να προσαρμόζουμε τις δράσεις για να πετύχουμε τα αποτελέσματα που θέλουμε. Τέλος πάντοτε θα παραμένουμε στις ε, δηλώσεις καλών προθέσεων χωρίς να μπορούμε να τους δώσουμε σάρκα και και να έχουμε χειροπιαστά αποτελέσματα. Προσοχή λοιπόν στο monitoring, στην παρακολούθηση και σε αυτό που καταφέρνουν τα προγράμματα να μας δώσουν βραχυπρόθεσμα. Ευχαριστώ. Κέλλη. Εκτός μικροφώνου. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω εκ των εισηγητή, τον κύριο Ντεμπάκερ για την ασιοδόξη του παρουσίαση και επιστημονική του παρουσίαση και για την καλή του δουλειά. Δύο πράγματα θα ήθελα να πω. Καταρχάς, όταν μιλάμε για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, μιλάμε για το μεγαλύτερο μέρος των επιχειρήσεων, πάνω από το 90%. Σχεδόν σε όλους λοιπόν ισχύουν, για όλους ισχύουν αυτά τα πράγματα. Κατά δεύτερον, θεωρώ ότι θα πρέπει να βάλουμε και ένα επίθετο, ε, εποφελής, ωφέλιμη κερδοφόρα πράσινη ανάπτυξη. Και όπως είπε και ο Πολ Ρουμπίκ, θα πρέπει να είμαστε πιο ανταγωνιστικοί στην Ευρώπη, να, να αναπτύξουμε την βιομηχανική μας βάση. Αυτό μπορούμε να το κάνουμε με πράσινο τρόπο και αυτό ακριβώς επισημαίνουμε. Και ιδιαίτερος πρέπει να κοιτάξουμε και το Κοινοβούλιο, το έργο του Κοινοβουλίου, αλλά και το έργο της Επιτροπής, όπου χρειάζεται κάποιες περιπτώσεις υποφελής αμοιβαία και για τη βιομηχανία, για παράδειγμα με τη μείωση αποβλήτων και απορριμμάτων, αν υπάρχει ανακύκλωση και αν είμαστε πιο αποτελεσματικοί σε ενεργειακά ζητήματα. Λοιπόν, κανείς δεν αντιλέγει ότι θα πρέπει να υπάρχει κερδοφορία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα αυτό και δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Θα πρέπει λοιπόν να το χρησιμοποιήσουμε αυτό, αλλά να συνδυάσουμε την ε, επικερδία, το κέρδος με την πράσινη ανάπτυξη, την προστασία του περιβάλλοντος και την ανάπτυξη βιομηχανικής βάσης και ανταγωνιστικότητα στον κόσμο. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε, αλλά ένα σκιώδης, ο κύριος Πιτικόφερ έχει το λόγο. Να σας ζητήσω συγγνώμη Πρόεδρε που άργησα. Ήμουν στο CDS. E Υποσχέθηκα όμως τον εισηγητή να τον υποστηρίξω και νομίζω ότι σε ό,τι αφορά τα θέματα αυτά είμαι αξιόπιστος. Which were... Ο Πρόεδρος, Ισκιώδης δεν τους περιμέναμε εδώ σήμερα το απόγευμα. Ποιος λοιπόν ήθελε να φύγει πρώτος, θα πρέπει να του δώσουμε το λόγο για την επόμενη έκθεση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό για μένα. Πολύ λυπάμαι που προσπαθώ να σας πιέσω χρονικά. Τώρα, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Κίρστη Έκροτ Μανσίλα. Έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και την ε, Επιτροπή σας. Πολύ χαίρομαι που άκουσα αυτά που είπατε και για την θερμή υποστήριξη του, του χάρτη πράσινης ανα, ε, ανάπτυξης. Χαίρομαι λοιπόν και ό,τι ιδέες έχετε θα ήθελα να τις ακούσω. Η Ευρώπη λοιπόν τώρα βρίσκεται σε μία οδό ανάκαμψης, χρειαζόμαστε ανάπτυξη και θέσεις εργασίες. Από που μπορούμε λοιπόν να τις βρούμε. Με την πράσινη ανάπτυξη είναι μια, έχουμε μία εξαιρετική ευκαιρία. Το μεγαλύτερο δυναμικό ανάπτυξης φαίνεται ότι προέρχεται από τις διατμήσεις μεταξύ των διαφόρων τομέων και από εκεί νομίζω ότι προέρχεται και πιο πολύ καινοτομία και σε ό,τι αφορά την κύκλικη οικονομία, εδώ θεωρώ ότι υπάρχει πολύ καλή δυνατότητα συνεργασίας. Εδώ λοιπόν υπάρχουν μεγάλες δυνατότητες ε, επιχειρηματικότητας. Όπως είπε και ο εισηγητής και οι συνεισηγητές, οι σκιώδεις, είναι μεγάλη η παγκόσμια αγορά και η Ευρώπη έχει μερίδιο 1 τρίτο σε αυτή την αγορά. Μόνο 10% εξαγωγές λοιπόν από μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Είναι τεράστιο το δυναμικό λοιπόν για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. κοιτώντα λοιπόν όλες τις ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, η αποτελεσματικότητα των πόρων μειώνει το κόστος παραγωγής και έτσι όλοι υποφελούνται στην διαδικασία παραγωγής. Είναι λοιπόν μια διπλά υποφελής κατάσταση για όλες τις εταιρείες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις κατά πάσα πιθανότητα γνωρίζουν λιγότερο από όλους ή έχουν το λιγότερο δυνατό χρόνο αν θέλετε από όλους για να αφιερώσουν σε αυτά τα πράγματα και με το σχέδιο δράσης. Λοιπόν, βρήκαμε 34 συγκεκριμένες δράσεις, μερικές εκ των οποίων έχουν να κάνουν πραγματικά με το τμήμα πληροφόρησης, ενημέρωσης, όπως το κέντρο αριστείας, για παράδειγμα, για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Έτσι, λοιπόν, ελπίζουμε να βελτιώσουμε τι αποδόσει των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και να διακρίνουν ποιε είναι οι επιχειρηματικές ευκαιρίες. Ε, προσβλέπουμε λοιπόν στην έκθεση και είμαστε ασφαλώ στη διάθεσή σα για ανταλλαγή απόψεων ή για ερωτήσει τι οποίε ενδεχομένω να έχετε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Να ζητήσω από του σκιώδει εισηγητέ αν έχουν κάτι να προσθέσουν. Μετά την παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κύριε Ρούμπι, κύριε Κόφορτ, Κύριε Ρούμπιχ. Βεβαίω, ο εισηγητή στο τέλο ε, για να ανακεφαλαίωση. Εννοείται. Ο κύριος Ρουμπίχ, είμαι και από την Επιτροπή ε, Προπολογισμού όπου και παρακολουθώ τη συζήτηση αυτή και το Συμβούλιο επιμένει για τις περικοπές των μέσων, όχι μόνο το πλαίσιο το έχει μειώσει κατά 4% μέχρι το 2020, αλλά και τον προπολογισμό ήτρε προσπαθεί όχι μόνο να μην δώσει τα παραπάνω χρήματα, αλλά να μην χρηματοδοτήσει και τα βασικά. Θα πρέπει να δούμε λοιπόν και να επικεντρωθούμε στις ε, εξαγωγές. Γι' αυτό λοιπόν να ζητήσω από την Επιτροπή να μας υποστηρίξει πλήρως, να μην επιτρέψουμε περικοπές προκειμένου το πρόγραμμα να διαμορφωθεί σε ένα πρόγραμμα πραγματική ανάπτυξη και να μπει στο επίκεντρο των προσπαθειών μα. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρο. Ο κύριο Ζόλο, εντάξει, πολύ ωραία. Ο εισηγητή. Να συνοψίσει παρακαλώ τι συζητήσει μα. Ε, Ευχαριστώ. Πρόεδρε. Ε, Συνοψίζοντα, θέλω να ευχαριστήσω όλου τους συνεργαστήκαμε μαζί για αυτήν την έκθεση και μέσα στο ίδιο μήκο κύματο, οπότε ε, ελπίζω να συνεχιστεί αυτή η καλή συνεργασία για να συνεχίσουμε. Κάτι άλλο το οποίο το είπε ο κ. Ρομπίχη. Να έχουμε κάποια εργαλεία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το Horizon 2020 και κάποια άλλα προγράμματα. Αλλά προσπαθώ να εστιάσω με την έκθεση το τι θα κάνουμε από πλευρά ιδιωτικών επενδύσεων. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό σε αυτήν την προβληματική. Να χρησιμοποιήσουμε τα ευρωπαϊκά χρήματα για να υποστηρίξουμε, να έχουμε ένα, ε, ένα πλαίσιο ε, καινοτομία στην αγορά. Η πρόκληση είναι πώς τα νέα προϊόντα θα μπουν στην αγορά, την ενιαία αγορά στην Ευρωπαϊκή. Ωραία να έχουμε νέες ιδέες, καινοτομία, νέα προϊόντα, αλλά τελικά θα πρέπει να φτάσουν εδώ στους καταναλωτέ. Άρα το θέμα είναι το πώς θα κόψουμε γραφειοκρατία. Να θέσουμε τα σχετικά προϊόντα στην εμπορία. Καλές είναι οι ιδέες που έρχονται και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Καλά τα νέα θα είναι στη διάθεσή μας. Ελπίζω ότι θα έχουμε ιδέες με τους επιχειρηματίες που θα συνομιλήσουμε πέραν των όσων αξιόλογων είπε η Επιτροπή. Και γι' αυτό και ελπίζω να έχουμε τελικά ε, μια καλή έκθεση που να αποτελέσει ένα ισχυρό μήνυμα προς τα έξω και προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο Πρόεδρος, σας ευχαριστούμε κύριε Σίγητα. Τώρα η συζήτηση της εκθέση θα γίνει 23 και 24 Δευτέρου του 2015. Δεν έχουμε τώρα το λεπτομερές πρόγραμμα των ημερών. Άρα ή 23 ή 24 θα ζητηθεί. Οπότε θα μας παρουσιάσει και το σχέδιο εκθέσεω ο συνάδελφος. Προθεσμία για υποβολή τροπολογιών. 25 Δευτέρου. Μία ημέρα μετά την συνεδρίαση της Επιτροπής. Αν το έχετε υπόψη. Τότε θα γίνει η συζήτηση. Και στις 25 θα λίγη προθεσμία που τροπολογιών Λέξανα πρώτος. Θέλουμε να έχουμε ολοκληρώσει πριν τις διακοπές. Και γι' αυτό θα πρέπει από τώρα να πούμε ότι η προθεσμία είναι 25 Φεβρουαρίου. Ξέρετε τι γίνεται. Χρειάζονται οι μεταφράσεις, δεν χρειάζεται να σας πω άλλα. Και τώρα συνάδελφοι, πάμε σε ένα άλλο επίσης σημαντικό ζήτημα της μεσής διατάξεως. Το αριθμός το παριθμό συγγνώμη, 11. Δημιουργία και λειτουργία αποθεματικού για τη σταθερότητα της αγοράς. Στον το σύστημα δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου και τροποποίηση της οδηγίας 2003. Κάθετο 87. Let me say that our rapporteur... Ο εισηγητής, ο κύριος Σταγιάννη, ενημερώθηκε ότι δεν θα αρχίσει μετά τις 4 παρατέταρτο η συνεδρίαση ή η συζήτηση του θέματός του μάλλον. Πριν από μισή ώρα το είπαμε. Όπου να είναι έρχεται. Είμαστε έτοιμοι να το συζητήσουμε. Το θέμα γιατί έχουμε το σχέδιο της ε, έκθεσης, έχουμε και τις τροπολογίες. Άρα μπορούμε να συζητήσουμε και τις τροπολογίες. Τα συζητήσαμε αυτά πάνω από μία φορά. Άρα μπορούμε να αρχίσουμε να το συζητούμε ε, και έχουμε τους ε, σκιώδεις ηγητές. Πρώτος ο κύριος Πίτερ Έριξον των Πρασίνων. Βιάζεστε, ξέρω. Ε, γιατί άλλαξε το πρόγραμμα και δεν ξέρω τι θα ζητηθεί το απόγευμα και όχι το πρωί. Ευχαριστώ. ήταν προγραμματισμένο για το πρωί. Και είναι καλό να προλάβω να πω αυτά που θέλω πριν φύγω. Η τελευταία, το τελευταίο θέμα που συζητήσαμε ήταν η πράσινη ανάπτυξη με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να πω ότι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο εδώ είναι να έχουμε σαφείς ξεκάθαρους στόχους για το μέλλον, για την βιωσιμότητα, καθώς και πολιτικά εργαλεία που να ανοίγουν το δρόμο για την βιωσιμότητα. Στην περίπτωση αυτή και με την κλιματική αλλαγή υπάρχουν εργαλεία για να αναχαιτήσουμε τις κλιματικές αυτές αλλαγές. Και το πιο χρήσιμο που έχουμε είναι το σύστημα εμπορίας εκπομπών. Η Επιτροπή έχει επικεντρωθεί σε ένα πραγματικό πρόβλημα σε αυτή την περίπτωση. Στο ότι το σύστημα ETS ε δεν λειτουργεί. Εδώ και καιρό δεν λειτουργεί Και καλό θα ήταν, ε, καλό είναι που ε, σκέφτεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λύσει αυτό το πρόβλημα με ένα αποθεματικό για τη σταθεροποίηση της αγοράς. Βεβαίως, ε, η προσπάθεια ήταν λίγο χλιαρή, διότι η Επιτροπή θα καθυστερήσει να προωθήσει το σύστημα αυτό και κάποιες από τις άδειες θα ε, περάσουν στο σύστημα του backload. Ε, θα πρέπει αυτά κάπως να τα αλλάξουμε. Ευτυχώς μπορέσαμε μεταξύ εισηγητών, ε, σκιωδών και κυρίως εισηγητή να τα δούμε αυτά. Και καλό θα να αναζητήσουμε την πλειοψηφία εφόσον όλα αυτά προχωρήσουν για να αλλάξει προς το καλύτερο η πρόταση της Επιτροπής. Ελπίζουμε να εγκριθεί και από το υπόλοιπο Κοινοβούλιο. Το πιο σημαντικό είναι ίσως να ξεκινήσει ο μηχανισμός αυτός, το αποθεματικό για τη του της αγοράς, MSR, να ξεκινήσει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα να λειτουργεί, ήδη από το 2017, και να ακυρώσουμε όλες τις άδειες που έχουν ε, υπολογιστεί προκαταβολικά στο σύστημα ή τέλο πάντων εκτό συστήματο πιο συγκεκριμένα. Και το τρίτο στοιχείο είναι ότι κάποιοι μιλάνε για τη διαρροή εκπομπών και συμφωνούν οι σκιώδεις ότι αυτό είναι λίγο εκτός πεδίου, θα πρέπει να επιληθεί σε άλλα σημεία, σε άλλα θέματα Α μην διαταράξουμε λοιπόν, ας διαταράξουμε το σύστημά μας και με αυτό το επιπλέον πρόβλημα. Και τέλος, υπάρχουν κάποιες ε, αλλαγές στις λεπτομέρειες. της πρόταση της Επιτροπής. Νομίζω ότι μπορούμε να συμφωνήσουμε στην Επιτροπή μας και να τα στείλουμε στην Ένβη έχοντας ήσυχη τη συνείδησή μας ότι κάναμε ό,τι μπορέσαμε για να φέρουμε τις σωστές αλλαγές και να λειτουργήσει επιτέλους το σύστημα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε Εκ μέρους του, των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, η κυρία Γκρίφιν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Συνάδελφοι, συγχαρητήρια για τη δουλειά σα σε αυτό το τόσο σημαντικό θέμα. Χαίρομαι που υπάρχει ευρεία συνένεση από τι πρώτε συναντήσει των εισηγητών μα και μεταξύ των διαφόρων πολιτικών ομάδων, σοσιαλιστών και δημοκρατών, γκουε, άλντε, για τα βασικά ε, θέματα του φακέλου αυτού. Θα πρέπει να ξεκινήσει νωρίτερα να λειτουργεί ο μηχανισμό για το αποθεματικό σταθερότητα τη αγορά, MSR, με άδειε που δεν θα πρέπει να επιστρέψουν στην αγορά, με υψηλότερα όρια και υψηλότερα ποσοστά για την απομάκρυνση αλλιών από την αγορά. Στην ίδια κατεύθυνση, Πρόεδρε, οδεύουμε για την ενίσχυση του συστήματο εμπορία εκπομπών με το MSR και με αυτήν την έκθεση ιδέα πρωτοβουλία. ως προς την ε, η ημερομηνία που προτείνουμε να είναι νωρίτερα, προτείνουμε το 2017 και ήθελα να κάνω κάποια σχόλια για τις τροπολογίες. Να υπογραμμίσω ότι δεν υπάρχει λόγος να περιμένουμε. Έχουμε ένα χαλασμένο εργαλείο και πρέπει να το φτιάξουμε όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Εάν προβλέψουμε το MSR το 2021, τα πλεονάσματα θα παραμείνουν υψηλά και τιμές χαμηλές. Οπότε το να στείλουμε λαθασμένα μηνύματα στους ενδεχόμενους επενδυτές των καθαρών τεχνολογιών για μια ολόκληρη δεκαετία ή παραπάνω δεν είναι η καταλληλότερη κίνηση. Επιπλέον δεν υπάρχει ε, σαφή συνένεση για την ε, αλλαγή της ημερομηνία. Υπάρχει, υπάρχουν κάποιοι που λένε ότι η βιομηχανία θα πιεστεί, ενώ κάποιοι άλλοι λένε ότι η βιομηχανία θα ωφεληθεί από μια σωστή τιμή για τις εκπομπές που θα οριστεί το Ένα μεγάλο μερίδιο επίσης του κλάδου ζητά όντως να προχωρήσει νωρίτερα η ημερομηνία θέση σε ισχύ. Επίσης υπάρχει απόφαση για το κατάλογο των τομέων που είναι εκτεθειμένοι στη διαρροή του άνθρακα έως το 2020. Για την ερχόμενη περίοδο τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Τόμπερ ε, υπογραμμίζουν και το παραθέτω ότι τα υφιστάμενα μέτρα θα συνεχίσουν μετά το 2020 για να προλάβουμε τον κίνδυνο της διαρροής άνθρακα. Αυτό δίνει τις απαραίτητες εγγύησεις μια πλειοψηφία χωρών στο Συμβούλιο πιέζουν επίσης για μια ε, αλλαγή της ημερομηνία και ο Επίτροπος Κανιέτε λέει ότι και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συμφωνήσει με την αλλαγή της ημερομηνία ε, θέση ίσχυ του MSR εφόσον συμφωνήσουν Συμβούλιο και Κοινοβούλιο. Το επιβεβαίωσε και χθε στην ακρόασή μας ε, όταν ρώτησα εάν θα μπορούσε να δεχτεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την ημερομηνία του 2017. Είναι λοιπόν ζωτική σημασία αυτή η ημερομηνία να συμπεριληφθεί στην γνωμοδότηση τη Επιτροπής μας. Επίσης ένα άλλο θέμα είναι αυτό που ανέφερε και ο συνάδελφος με το backload των αδειών. Εδώ ε, θα πρέπει να ακυρώσουμε τις άδειες αυτές οι οποίες θα έρθουν πάλι στην αγορά το 2019. Το να φέρουμε 900 εκατομμύρια ε, άδειες ε, καθυστερημένες στην αγορά θα ήταν παράλογο και θα δημιουργήσει τριγμούς και στρέβλωση. Ως προς τα επιτόκια τα ποσοστά μάλλον, ο στόχος μας είναι να, ε, να ενισχύσουμε το MSR και να είναι ένα ε, επιτυχημένο ε, εργαλείο. Γι' αυτό τα ποσοστά από, κράτη, από μάκρυσης πρέπει να είναι στο 20% και η υπερβολική παροχή προς την αγορά μπορεί έτσι να εξαλειφθεί στο 2024. Επίσης το το όριο πρέπει να, κατα... να φτάσει τα 300 εκατομμύρια με εκατότατο όριο που θα αποτρέπει την υπερβολική ε, πάροχη προς την αγορά που είναι τώρα το μεγαλύτερο ζήτημα. Και τώρα προς τη διαρροή του άνθρακα, Πρόεδρε, θα πρέπει να υπάρχει ένας εύχριστος κατάλογος για τη διαρροή του άνθρακα με τα σωστά κίνητρα. Κατά τρίτον, πιστεύω ότι αυτή η γνωμοδότηση για το ε, σύστημα, για το αποθεματικό σταθερό της αγοράς, εδώ μιλάμε για τον όγκο αδειών που θα υπάρχουν στην αγορά και όχι για τις δωρεάν αδειές που θα δοθούν στην ε, βιομηχανία. Επίσης δεν υπάρχουν αποτελέσματα για το πόσο διαρροή άνθρακα υπάρχει εξαιτία του συστήματος εμπορίας εκπομπών. Την διαρροή του άνθρακα πρέπει να αντιμετωπίσουμε στο 2020 και υπάρχουν σχετικά μέτρα. Ε, ο κλάδος μαζί με όλους που θα μπορούσαν να αποφεληθούν από την μεταρρύθμιση του συστήματος ETS στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, πιέζει και θα πρέπει αυτό να ληφθεί υπόψη και από τον εισηγητή στις συμβαστικές του προτάσεις. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Ισηγητά, κύριε Αντιπρόεδρε, ξεκινήσαμε γιατί βιάζονται οι σκιώδεις μας και επίσης ε, βιάζεται πολύ και κύριο Πέντελε. Αν θα μπορούσατε να κάνετε τώρα την παρέμβασή σας. Κοιτάξτε. Ο κύριος Τατζάνη μπορεί να πάρει το λόγο πριν από μένα. Δεν βιάζομαι, δεν βιάζομαι, λέει ο κύριος Μάλιστα, πολύ ωραία. Λυπάμαι σκιώδες εισηγητές για την αλλαγή αυτή που έγινε στο χρονοδιάγραμμα. Οι δύο σκιώδες, κύριε Σκρομπάτσο και κυρία Ένστου, δεν είναι εδώ μαζί μας σήμερα γιατί ήταν αδύνατο να μείνουν παραπάνω. Ίσως την επόμενη περίσταση. Ε, επειδή σε κάποιες περιπτώσεις ο εισηγητής μας δεν μπορεί να είναι παρόν. Το καταλαβαίνουμε στην περίπτωση αυτή ο συντονιστής από την ίδια πολιτική ομάδα θα μπορούσε να κάνει κάποιες εισαγωγικές ε, παρατηρήσεις ε, εξ ονόματος του εισηγητή και να παρουσιάσει το θέμα αυτό στον εισηγητή γιατί σήμερα μας λείπουν ε, δύο σκιώτες οι οποίοι ήταν από το πρωί. And Mr. Ο κύριος εισηγητής λοιπόν, ο κύριος αντιπρόεδρος έχει το λόγο. Έχετε το λόγο. Σας... Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Να σας πω πως έχει κατάσταση μετά τη συνάντηση πριν από ένα 15 θήμερος για αυτή την έκθεση. Ξέρετε ποια είναι η θέση μου, παραμένει η ίδια. Και προχθές συναντηθήκαμε όλοι με τους πιο δυσηγητές και θέλω να τους ευχαριστήσω γιατί συνέβαλαν και την ε, Παρασκευή υποβλήθηκαν οι τροπολογίες για το κείμενο είναι κάτι παραπάνω από 100 και επικεντρώνεται σε πέντε βασικά θέματα. Το πότε θα αρχίσει να ισχύει ο μηχανισμός MSR. Όλοι θέλουν να γίνει αυτό λίγο, λίγο πιο νωρί, άλλοι πιο αργά. Επομένω, εγώ δεν θα αλλάξω την αρχική πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή που έλεγε να ξεκινήσει αυτό στις, το 2021. Και σύμφωνα η δεύτερη ομάδα αφορά τα, τα, τα, τα κατόφλια για τα οποία θα πρέπει να μπουν στο, αυτό στο, στο αποθεματικό για σταθερότητα και μερικοί θέλουν να είναι πιο ψηλό, άλλοι πιο χαμηλό. Αυτό το κατόφλι, εγώ λέω, να είναι στο 12 με 15% τρίτη ομάδα είναι το backlog. Και η πρόταση της Ευρωπαϊκής δεν έλεγε ποιες θα, θα, είναι, αυτές οι άδειε. Και λέμε ότι αυτό πρόκειται να ανακατέψει την αγορά και είπαμε ότι αυτό θα γίνει 2019-2020. Και τώρα η τέταρτη ομάδα των τροπολογιών που θα πρέπει να αφορά την διαρροή για να προστατεύσουμε τη βιομηχανία. Οπότε νομίζω ότι Έχουμε εδώ πέρα περίπου την κατάσταση και είπαμε ότι έχουμε την οδηγία ETS για τις εκπομπέ. και αυτό αφορά έναν μηχανισμό και επομένω χρειάζεται να δούμε πότε θα ξεκινήσει η αγορά και αυτό θα το εξετάσουμε για να δούμε αν αυτό λειτουργεί ή όχι. Η Επιτροπή είναι διαθέσιμη και θέλει να γίνει η αναθεώρηση της οδηγίας όταν ε, ε, εγκριθεί αυτός ο MSR και για μένα αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Δεν θέλω να επαναλάβω τα ίδια για αυτό το επιχείρημα, αλλά νομίζω ότι είναι σημαντικό η Επιτροπή να υπεραμεινθεί της Ευρωπαϊκής Βιομηχανίας, ούτως ώστε το τελικό κείμενο να είναι ισορροπημένο σε σχέση με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. ε, είμαι αισιόδοξο, οπότε θα ήθελα να καταλήξουμε με κάποια ε, λύση συνενετική με όλους εμπλεκομένους στην Επιτροπή. Και τώρα πρότεινα κύριε Πρόεδρε ε, με τους δύο συγγητές να δούμε πρώτα-πρώτα κάποιες ε, ε, ε, συμβαστικέ τοπολογίε στι 8 12 και σε μια δεύτερη συνάντηση με του κοινοδοσηγητές να τα να ξαναδούμε οριστικά στο Στρασβούργο την επόμενη εβδομάδα να συναντηθούμε να δούμε πώς συμφωνήσουμε με τους οι συνεργάτες μας και να μπορούμε να δούμε πώς έχουν τα πράγματα και κατόπιν να συναντηθούμε στο Στρασβούργο όπου να καλέσουμε και τον Ιβο Μπέλε της Ένβη και έτσι να δουλέψουμε μαζί. Και ο μπέλετ τόσα χρόνια ήταν σε αυτή την επιτροπή και παρακολουθεί με ενδιαφέροντα Εδώ εδώ τεκτενόμενα, οπότε εάν σύμφωνη τον... να τον ε, καλέσουμε σε αυτή τη συνεδρία στο Στασβούργο. Και μετά, πριν την ε, ψηφοφορία, να συναντηθούμε τον Ιανουάριο Συγγνώμη που καθυστέρησα και που έτσι συζητήσαμε την έκθεση λίγο πιο αργά. Ευχαριστώ πολύ ο Πρόεδρος. Είναι πολύ καλό που είναι εδώ και ο συνάδελφος Μπέλετ, οπότε μπορούμε να τα συζητήσουμε και μαζί σας. Όμως θα ζητήσω από τον κύριο Γκουμπάρτσικ να πάρει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Βεβαίως, να πω και εγώ μερικά για αυτό το θέμα. Συμφωνούμε με έννοια και την προσέγγιση του κυρίου Ταγιάννη με την ε, συλλογιστική που προτείνει, όμως υπάρχουν κάποια σχόλια για τα βασικά ζητήματα από πλευράς μας. Λόγω χάρη η Προθεσμία. Είναι κάπως νωρίς δεδομένη στις κρίσεις στην Ευρώπη και τις απειλές προς την ευρωπαϊκή οικονομία. Για μας σημαντικότερο είναι να προστατεύσουμε τη βιομηχανία, κάτι που το έθιξε ο κ. Σταγιάννη βέβαια, αλλά και να προστατεύσουμε τις θέσεις εργασίας. Νομίζω ότι δεν είναι καλή ιδέα να δημιουργήσουμε προβλήματα με ένα πρόχειρα φτιαγμένο σύστημα και με την ανακατανομή των δικαιωμάτων. Κάποια από τα δικαιώματα έχουν ε, αποσυρθεί από την αγορά. Οπότε πρέπει να τα μέτρα που θα λάβουμε να προστατεύουν τον κλάδο αυτό. Δεν μπορούμε να έχουμε λίγα πιστοποιητικά ε, που να λίγες άδειες που να κυκλοφορούν στην αγορά, γιατί έτσι θα αυξηθούν πολλοί τιμέ απότομα και θα έχουμε πάλι πρόβλημα. Θα πλήξουμε την βιομηχανία, το σχετικό κλάδο και πιστεύουμε ότι αυτός θα πρέπει να είναι το πρώτο μα μέλημα. Ω προ την αναθεώρηση, πιστεύουμε ότι η τριετία είναι πολύ μεγάλο διάστημα. Θα πρέπει να το μειώσουμε στον ένα χρόνο και να ε, επανεξετάσουμε την κατάσταση μετά το πέρας ενός έτους ώστε να αντιμετωπίσουμε τις τρευλώσει που μπορούν να προκύψουν στην αγορά σχετικά. Ευχαριστούμε. Κύριε Φέντερλι. Ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ και τον κύριο Ταγιάννη για την έκθεση του. Νομίζω έγινε σαφές όταν είδαμε τις τροπολογίες ότι έτσι κι αλλιώς δεν ήταν όλες μεταφρασμένες στα αγγλικά, οπότε κάποιες δεν τις έχουμε διαβάσει ακόμα, όμως αυτές που μπορέσαμε να διαβάσουμε από τη συνάντηση των σχεδόν της προάλλες, φαίνεται να δείχνουν ότι όλοι σχεδόν από το σώμα μας θέλουν την μετακίνηση της ημερομηνία το 2017. Και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ακούμε τέτοιες ειδήσει, εάν το επιθυμήσουμε και εμείς και το Συμβούλιο. Εάν σωστά τα έχω σημειώσει, η ALDE, η ΣΝΤ, η GUE και ε, οι Σοσιαλιστές και οι Δημοκράτες, μέρη του ΕΛΚ και μέρη των συντηρητικών και μεταρρυθμιστών είναι υπέρ της ημερομηνία αυτής. Με 11 χώρες τουλάχιστον να είναι επίσης υπέρ στο Συμβούλιο θα πρέπει να προστατεύσουμε τους κλάδους. Δεν μπορούμε να τους λέμε ότι θα είναι τόσο εξευτελιστικά χαμηλές όπως τώρα για πάντα. Η πολύ χαμηλή τιμή των δικαιωμάτων εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου θα οδηγήσουν σε λάθος σε λάθο είδου επενδύσεις. Και αυτό πρέπει να το δούμε και το, πριν το 2020, διότι ο κλάδος θα μας πει ότι είναι πολύ φτηνέ τιμέ επί τόσο καιρό και ξαφνικά ε, ακρίβηναν και ανέβηκαν τόσο τιμέ. Δεν το είπατε πριν από τόσα χρόνια ε, ο κλάδος θα χάσει την εμπιστοσύνη του. Ε, στοχεύει σε υψηλότερε τιμέ ο κλάδο ε, για τις ανταλλαγέ. Επίσης δεν πιστεύω ότι τα δικαιώματα που είναι αντικείμενο του backlog θα πρέπει να επιστρέψουν στην αγορά. Βλέπω να λέει ο κ. Σταγιάννη ότι θα μπορούσαν ε, να μπουν στο αποθεματικό προσωρινά. Δεν τις ε, αποσύρουμε τελείως έτσι, δεν τις εξαλείφουμε, αλλά η εξάλληψή τους ε, θα είναι μοιραία αργά γρήγορα, γιατί δεν βοηθούν κανένα. Μπορούμε λοιπόν είτε να τις ακυρώσουμε αμέσως, είτε να τις βάλουμε στο αποθεματικό και να καθυστερήσουμε την κατάργησή τους, την ακύρωση ολοκλήρωση των δικαιωμάτων αυτών που είναι αντικείμενο backlog. Μπορούμε να το συμφωνήσουμε μεταξύ μα. Όμω βλέπω ότι είναι πολλά τα μέλη του ε, Κοινοβουλίου που ε, θέλουν να αποσταλεί ένα ισχυρό μήνυμα και προ την Επιτροπή και προ το Συμβούλιο. Ε, είμαι κατά ιασδήποτε μνήμα στη διαρροή άνθρακα και ένα σχετικό κατάλογο. Αυτό θα το δούμε εν ευθέτω χρόνο, θα υπάρξει αναθεώρηση σε λίγα χρόνια, αλλά νομίζω ότι προσπαθούμε να ότι θα το υποβαθμίσουμε το θέμα και μάλιστα δει εφόσον το συμπεριλάβουμε από το κείμενο. Ε, έχουν γίνει απαραίτητε αλλαγέ όταν ε, εγκρίθηκε το 2003. Εάν λοιπόν τη συζήτηση για τη διαρροή του άνθρακα τη μετακινήσουμε στην έκθεση αυτή, ε, θα περάσουν πράγματα που δεν θέλουμε μέσα από το Κοινοβούλιο. Τώρα πρέπει να δώσουμε σταθερότητα στην αγορά, πρέπει να υπάρξει μια σύντομη αναθεώρηση για να δούμε αν τα στοιχεία που συμφωνήσαμε ήταν τα σωστά και αν μπορούν να επικρατήσουν για περισσότερο καιρό. Θα ήθελα αυστηρότερα όρια και όταν είδα τις τροπολογίες πρόσεξα ότι κάποιοι θέλαν χαλαρότερα όρια. Όμω η συντριπτική πλειοψηφία, για να αρχίσουμε πάλι να, μιλά να μετράμε πολιτικέ ομάδε, οι περισσότεροι στο Κοινοβούλιο είναι υπέρ τη μεγαλύτερη αυστηρότητα στα όρια. Θα υποβάλλω τροπολογίε για χαμηλότερου αριθμού αριθμούς στα κατόφλια, τις οροφές και τους αριθμούς και θα έλεγα ότι θα πρέπει περισσότερες άδειες θα πρέπει να έχουν δικαίωμα πρόσβαση στο αποθεματικό. Έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας και Θέλουμε το σύστημα αυτό να αρχίσει να λειτουργεί γρήγορα, εάν επιθυμούμε ισχυρή πράσινη οικονομία στην Ευρώπη, αλλά και έναν βιώσιμο τρόπο για τη βιομηχανία μας να λειτουργεί. Η συζήτηση στο Κοινοβούλιο πρέπει να αποφασίσει εάν θέλουμε να συνεχίσουν να λειτουργούν ως έχουν οι εταιρείε ή αν θέλουμε να τι προσελκύσουμε στην αγορά για να δημιουργήσουν νέες θέσει εργασία. Νομίζω ότι η λύση μα είναι η δεύτερη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε εκ μέρους των φιλελευθέρων. Μιλήσατε. Τώρα η κυρία Ένστ, εκ μέρους της Γκουε. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και τον εισηγητή. Θα ήθελα να του πω ότι ήταν πάρα πολύ καλό να συμφωνήσουμε επί των απόψεών μας στις συναντήσεις των σκιωδών και η δικιά μας ομάδα προφανώς έχει διάφορα σημεία τα οποία επικρίνει να σας πω ότι δεν είμαστε υπέρμαχοι του εμπορίου ρήπου. Νομίζω ότι αυτό είναι γνωστό άλλωστε. Αλλά ασφαλώς θα πρέπει με ρεαλιστικό τρόπο να αντιμετωπίσουμε την πρόταση, το οποίο και πράξαμε. Ε, κάναμε δύο προτάσεις, ε, αλλά είμαστε και ρεαλιστές, είμαστε πραγματιστές, γι' αυτό λοιπόν θα θέλαμε να ακολουθήσουμε την εξής πρόταση. Τα πιστοποιητικά στην πρώτη φάση των τριών ετών θεωρούμε ότι δεν φτάνουν. Θα πρέπει να έχουμε πιο πολλά πιστοποιητικά. Αυτό λοιπόν είναι το πρώτο σημείο. Αυτό που δεν θέλουμε, είτε πρόκειται για 900 εκατομμύρια, είναι να μην επανέρχεται το ποσό αυτό στην αγορά. Αυτό το είπαν διάφοροι, εμένουμε σε αυτό. Ιδάλλως θεωρούμε ότι δεν υπάρχει καμία επίδραση στο σύστημα αυτό. Το επόμενο σημείο που ήθελα να θίξω έχει να κάνει με το άρθρο 3, σημείο 3. Συγγνώμη, άρθρο 1, σημείο 3. Για το έτος 2021 ε, θεωρούμε ότι είναι πολύ αργά. Πιστεύουμε ότι θα πρέπει να βρούμε μια πιο νωρίς ημερομηνία για το 2015, το οποίο το συζητούν και άλλες ομάδες. Τώρα, επίσης για το 12% κατά πόσον αρκεί αυτό για τη συνολική ποσότητα, αμφιβάλλουμε. Θεωρώ ότι θα πρέπει να είναι παραπάνω το ποσοστό αυτό, αλλά αυτό μπορούμε να το διαπραγματευτούμε. Τέταρτο σημείο αφορά τα πιστοποιητικά που κυκλοφορούν Αντί 400 εκατομμύρια θα θέλαμε 500, 600 εκατομμύρια. Και αυτό μπορούμε να το συζητήσουμε και θα πρέπει να το συζητήσουμε ενδεχομένω με τις τροπολογίες να το αλλάξουμε. Σε ό,τι αφορά τη συζήτηση για τη διαρροή άνθρακα, θεωρούμε ότι δεν προχωράει η συζήτηση και θα θέλαμε λοιπόν ε, να απομακρυνθούμε από τη συζήτηση και έτσι λοιπόν υποστηρίζουμε πολλούς από αυτούς που πήραν το λόγο για το θέμα αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρος. Αν μου επιτρέπετε να ζητήσω από την κυρία Γκρίφιν, θέλει να προσθέσει κάτι όσο είναι εδώ ο εισηγητής. Αλλά αν θα θέλετε παρακαλώ μη μακρηγορήσετε ένα λεπτό και λυπάμαι αν σας περιορίζω. Όχι καθόλου πρόεδρε, δεν πειράζει. Αγαπητέ εισηγητά. Τα σημεία που αναφέραμε, όπως είπε ο συνάδελφος, ε, υπάρχει μεγάλη ευρεία συνένεση, μάλλον που ε, ανακύπτει μεταξύ σοσιαλιστών, γκουε και πρασίνων και άλλα συγγνώμη για το MSR για το 2017 για τις, ε, το backloading που δεν θα πρέπει να επιστρέψει στην αγορά μεγαλύτερο ποσοστό αδειών από την αγορά και να ενισχύσουμε τη σχέση με το MSR. Αυτά θα θέλαμε λοιπόν να ληφθούν υπόψη στο σχέδιο γνωματότησης. Προτείνουμε το 2017 γιατί δεν έχει λογική το να περιμένουμε. Αν υπάρχει ένα μέσο το οποίο δεν λειτουργεί, ας το διορθώσουμε το συντομότερα δυνατόν. Θα γνωρίζετε ότι χθε στην Επιτροπή μας ο κ. Κανέτα είπε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα υποστηρίζει σε πρώιμη φάση, νωρίτερη φάση, το MSR αν επιβεβαίωνε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Γι' αυτό λοιπόν είναι κρίσιμο να συμπεριληφθεί μια πιο πρώιμη ημερομηνία και σε ό,τι αφορά το backloading, όπως είπαν οι συνάδελφοι, για το θέμα της διαρροής αερίου. Υποστηρίζουμε μια καλή λίστα, αλλά το MSR είναι κάτι διαφορετικό. Έχει να κάνει με την ποσότητα των αδειών και όχι με τις ίδιες άδειες που δοθούν στην βιομηχανία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λέει ο Πρόεδρος, να ρωτήσω λοιπόν από τον Ιβο ε, Μπέλε, το οποίο είναι πρώην πλήρες μέλος της Επιτροπής Ήτρε, να μας παρουσιάσει τη δική του έκταση, που είναι και η πιο σημαντική για μας. Όπως είπε και ο συγγητής κ. Σταγιάννη, θα σας στείλουμε κάποιες κρίσιμες ε, γνωμοδοτήσεις. Συγγνώμη σας, λοιπόν, έχει ιδιαίτερο βάρος. Γιάννη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Όχι, δεν ήταν χρόνια. Πριν από λίγους μήνες απεχώρησα από την Επιτροπή σας. Όντως, ο χρόνος περνάει πολύ γρήγορα και εδώ γύρω μου βλέπω τόσα ειδική πρόσωπα. Χαίρομαι που ήρθα εδώ και ευχαριστώ που μου δώσατε το λόγο και με μεγάλο ενδιαφέρον διάβασα τις άνω των 100 τροπολογίες του, για την οπότε τα περισσότερα τα ακούσατε, αλλά εν συνόψη να πούμε ότι υπάρχει μια πλατφόρμα συνένεσης, ώστε το σύστημα ανταλλαγών να μεταρρυθμιστεί και να έχουμε και το ταμείο αυτό για την σταθερότητα. Έχουμε την πρώτη τροπολογία, την υπέβαλαν δύο ή τρεις και ζητούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αποσύρει την πρόταση. Αλλά νομίζω ότι αυτό είναι καθαρά μειονοτική άποψη, γιατί οι περισσότεροι θέλουν να υπάρξει μεταρρύθμιση φοβούνται ότι το ETS θα καταρρεύσει. Όχι από τα 30, από τα 7 ευρώ που είναι τώρα. Ε, η τιμή και θα πάει ακόμα χαμηλότερα. Οπότε η συζήτηση όλη αφορά τις λεπτομέρειες της ε, μεταρρύθμισης και περιμένω τις ε, συμβαστικές προτάσεις που θα υποβάλει στο άμεσο μέλλον ο κ. Σταγιάννη από τα βασικότερα στοιχεία είναι αυτά τα 900 εκατομμύρια το πειράξαν να πέσουν στην αγορά. Αποφασίσαμε για το 2019 και το 2020 και νομίζω συμφωνούμε και στις δύο επιτροπές ότι αυτό είναι μια λογική λύση. Να μην μπουν στην αγορά και με το MSR να ξαναπάνε στο αποθεματικό. Δεν θα ήταν καλό αυτό, θα δημιουργούσε ακόμα ένα σοκ στην αγορά και κανείς δεν θέλει κάτι τέτοιο. Οπότε δεν ξέρω αν πρέπει να ματιωθεί αυτό. Εγώ πρότεινα όλα αυτά να μεταφερθούν στο αποθεματικό, λιγότερο ριζοσπαστικό. Και άκουσα τον κύριο Φέντερλε ότι τι λέει, είπε για late kill, δημιουργικός, γλωσσοπλάστης. Να το δούμε. Αυτό το, αυτό το, το late kill, το, το, βολή που έρχεται στο τέλος. Κάπως έτσι. Λοιπόν, για να δούμε τώρα τι γίνεται με το άνω κατόφλι, το κάτω κατόφλι τα 400 εκατομμύρια ή την άλλη πόλη τα 500 πόσα είναι. Οπότε να δούμε τι γίνεται και με τις δύο κατευθύνσεις, προς το ανέβασμα και προς τα κάτω, προς την ευελιξία. Εγώ έχω προτείνει να μην αγγίξουμε αυτά τα κατόφλια, να τα αφήσουμε όσοι είναι, να μείνουμε στην πρόταση της Κομισιόν. Δεν ήρθαν εδώ, θα έρθουν μετά, αλλά τέλος πάντων. Να το συνδυάσουμε με κάποια αναθεώρηση πρώτερη όπως είπατε και να γίνει αυτό ταχαίως αν γίνεται μετά από ένα χρόνο ο κ. Γκαρμπάτσης και είπε κάτι για ένα χρόνο ε, αυτό παρά είναι νωρίς δεν ξέρω αν η Κομισιόν μπορεί να το κάνει αυτό μόλις μετά από ένα χρόνο καλά μπορεί να, το βρούμε κάπου στη μέση Τώρα το θέμα της διαρροής. Κύριε Γκρίφιν, σωστά άκουσα την καταλαβαίνω. Τι είπατε ότι δεν είναι ήρθε τώρα η ώρα εδώ δεν είναι ο σωστό τόπος στο νομοθέτημα αυτό να ρυθμιστεί. Αλλά ε, κάπως διαφωνώ όσον αφορά το ότι πρέπει να δώσουμε το μήνυμα. Να στείλουμε το μήνυμα εδώ και η NVK Ήτρε προς Κομισιόν και Συμβούλιο για να του πούμε ότι θέλουμε να είναι ξεκάθαρο το μήνυμα ότι συμμεριζόμαστε τις ανησυχίες της βιομηχανίας ότι υπάρχει κίνδυνος διαρροής, ακόμα και πριν το 2020, σίγουρα μετά. Επομένως, σαφές μήνυμα στην Κομισιόν ότι θα πρέπει το συντομότερο να υπάρχει μια πρόταση μεταρρύθμισης, μόλις αυτή εγκρίθηκε. Αν όχι μετά από ένα-δύο χρόνια, άντε έξι μήνες μετά την επίσημη πρόταση, να συμβαστούμε για το πότε, να μην προσπαθήσουμε τώρα επομένως να το ρυθμίσουμε, αλλά να στείλουμε το, σήμα, το μήνυμα προς τους ε, εταίρους μας τα άλλα θεσμικά όργανα. Αυτά είναι τα πιο σημαντικά σημεία, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, ευχαριστώ, λέει Ευχαριστώ. Ρούμπικ. Äh, Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Νομίζω ότι αυτό που χρειάζεται βιομηχανία είναι και μια αξιόπιστη νομοθεσία. Δεν είναι λοιπόν ε, σωστό και καλό κάθε χρόνο να εξετάζουμε την ομοθεσία και πρώτα και γεγονός ότι υπάρχουν στόχοι για το 2020 διαρκώς να προσαρμόζονται. Η βιομηχανία λοιπόν πρέπει να επενδύσει και κάνει, λαμβάνει αποφάσεις για τις επενδύσεις. Οι αποφάσεις αυτές έχουν 50 χρόνια διάρκεια. Αν λοιπόν διαρκώς αλλάζουμε τη στοχοθεσία είναι πάρα πολύ δύσκολο να επενδύσουν σωστά και από την άλλη έχουμε και μια μεγάλη ανεργία και παρά το γεγονός ότι έχουμε τις πιο βιώσιμες μηχανίες στον κόσμο είναι τόσο δυναμική η νομοθεσία και αποτελεσματική που είναι δύσκολο να την παρακολουθήσει κανείς και είναι δύσκολο κανείς να προβλέψει πώς θα εφαρμοστούν όλα αυτά στο μέλλον. Ξέρουμε ότι και η οικονομική πολιτική, η χρηματοπιστωτική πολιτική δραματίζει πλέον σημαντικό ρόλο και όσα έχουν να κάνουν με τα παράγωγα που υπάρχουν εδώ. Υπάρχει διπλή επιβάρυνση με την παραγωγή της ενέργειας και κατά δεύτερον όταν καταναλώνεται αυτή η ενέργεια στην παραγωγή προϊόντων. Είναι διπλό λοιπόν αυτή η επιβάρυνση και πολύ απλά πρέπει να αναρωτηθούμε πώς θα προχωρήσουμε στο μέλλον σε ό,τι αφορά το θέμα της διαρροής. Θα πρέπει να σταματήσουν να υπάρχουν αυτές οι διπλές επιβαρύνσεις. Γιατί πραγματικά θα πρέπει να υπάρχει σταθερή νομοθεσία. Δεν υπάρχει καμία, κανένα πρόβλημα να συζητήσουμε ξανά τα θέματα για τους στόχους του 2020 και να θέσουμε καινούργιους στόχους για το 2030, αλλά να κάνουμε μελέτη αντικτύπου το συντομότερο δυνατόν για να δούμε τι σημαίνει αυτό για τις θέσεις απασχόλησης. Θα μπορέσουμε πραγματικά με τις νέες αυτές τις προτάσεις να δημιουργήσουμε νέες θέσεις εργασίας, καλοπληρωμένες ή μήπως θα καταστρέφουμε όλα. Γιατί αν δεν είναι σίγουρο ότι θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας, θα πρέπει να σκεφτούμε το όλο σύστημα. Θα πρέπει βιώσιμα λοιπόν εφαρμοστούν όλα αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Συνάδελφο Κέλλη. Εκτός μικροφώνου. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Νομίζω ότι μπορούμε να φτάσουμε σε ικανοποιητικές συμφωνίες για το θέμα αυτό με τη συνεργασία του πρώην Επιτροπού Ταγιάννη και του κυρίου Μπέλετ και που είναι ακόμα μαζί μας να πω ότι οι τροπολογίες 24, 40 και 73 δεν έχουν ακόμη συμπεριληφθεί στο κατάλογο. Ελπίζω να προσθεθούν, ιδίω για την 73. Νομίζω ότι όντω πρέπει η ημερομηνία να αλλάξει από 2021 σε 2017. Όλοι συμφωνούμε ότι θα έχει περισσότερο νόημα και επίσης να υπάρξει μια ημερομηνία και για την αναθεώρηση που προβλέπεται 2022 ας πούμε όπως προτάθηκε αρχικά είναι ίσως πολύ αργά. Αυτή ήταν η δική μου συνεισφορά. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε ο Χόκμαρκ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Άκουσα τη συζήτηση και μία σκέψη μου έρχεται στο μυαλό. Ο στόχος μας δεν είναι να δημιουργήσουμε το τέλειο σύστημα απομονώνοντάς το από την πραγματικότητα. Κάποιες φορές όταν ε, αμολάει κανείς τους πολιτικούς, τους θεωρητικούς, τους πολιτικούς ευθύνονται σε ένα θέμα, τείνουν να μην μαζεύονται. Όμως δεν είναι αυτό το πρόβλημά μας. Θέλουμε να δημιουργηθεί ένα σύστημα που να διευκολύνει τον ε, σχετικό κλάδο να αναπτυχθεί στην Ευρώπη. Να συμβάλλουμε στην ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας ενώ εμείς θα πετύχουμε ταυτόχρονα το στόχο μείωσης των αερίων του θεραποκηπίου της μείωσης ρήπων διοξιδίου του άνθρακα να θυμηθούμε ότι οι στόχοι αυτοί συνδυάζονται και με ένα σωρό άλλους τομείς και πολιτικές στη φορολογία, άλλους κανόνες των κρατών μελών που επιδιώκουν τον ίδιο στόχο. Δεν είναι αυτό το μόνο όργανο που διαθέτουμε. για να επιδιώξουμε τον ίδιο στόχο. Απλώς κάποιες φορές έχω την αίσθηση ότι κάποιοι θέλουν να χρησιμοποιήσουν αυτό σε πρόσχημα για να επιδοτήσουν τον κλάδο ή για να τον τιμωρήσουν. Ε, και δεν είναι αυτός ο στόχος μας, είναι να δημιουργεί ένα σταθερό, ένα σαφές πλαίσιο για να βοηθήσουμε τον κλάδο και να πετύχουμε πραγματικές μειώσεις. Νομίζω ότι πρέπει να είμαστε εδώ πραγματιστές και ρεαλιστές. Μην επιδιώκουμε το τέλειο σύστημα, όπως όταν παίζαμε με τα κουκλάκια, με τα σπίτια ε, από κούκλες ή τα κουρδιστά αυτοκινητάκια όταν ήμασταν παιδιά, κοριτσάκια και αγοράκια διότι αυτό το λέω πολύ σοβαρά και τη συζήτηση αυτή την ε, έχω κάνει και στη Σουηδία. Μερικοί παθαίνουν αιμονή. Όχι, μιλάμε για το μέρος ενός, ενός ολοκληρωμένου πλαισίου για τη μείωση των ε, αερίων διοξιδίου του άνθρακα. Ευχαριστούμε ο κύριος Ταμπουράνο. Εγώ προέρχομαι από έναν κλάδο, τον ιατρικό κλάδο. Και πολλές φορές διαλέγουμε μια θεραπεία ως γιατρή, την πιο αποτελεσματική για το σκοπό. Εάν διαπιστώσουμε ότι δεν λειτουργεί και δεν αλλάζουμε τη θεραπεία, αυτό σημαίνει ότι είμαστε κακοί γιατροί. Το ETS ίσως δεν είναι η καλύτερη μέθοδος. Ίσως έπρεπε να διαλέξουμε άλλη λύση για το πρόβλημα των εκπομπών. Ακόμα και αυτό το, το, το, βρήκαμε τότε που δεν είχαμε τέτοια παγκοσμιοποίηση. Ίσως θα πρέπει να κάνουμε επιμένως κάτι τελείως διαφορετικό. Δεν συμφωνούμε όσον αυτό ότι πρέπει να φέρουμε πιο μπροστά τη θέση σε ισχύ του μηχανισμού σταθερότητας του, ταμείου αυτού. Ίσως πρέπει να το σκεφτούμε καλύτερα. Αφού λοιπόν ένα σύστημα δεν έχει αποδώσει. Θέλουμε να κάνουμε το back London και τώρα θέλουμε να κάνουμε αυτό το αποθεματικό σε σχέση με την, με κατάσταση αυτών, τη μεταφορά τους αυτών των ποσοστώσεων. Δεν θα γίνει τίποτα για τις εκπομπές παγκοσμίω. Ούτε βέβαια θα βοηθήσει την βιομηχανία. Ούτε πρόκειται να έχουμε τώρα κάποιες βιομηχανικές πρακτικές με λιγότερες εκπομπές. Θα πρέπει κάποια ομάδα εργασίας να κάτσουμε και να βρούμε ένα καινούριο σύστημα. Έναν ε, φόρο carbon tax που να μην αναλογεί στην αγορά αλλά να έχει κάποιο είδου ε, μεταβλητές θερμοδυναμικής και κάτι το οποίο να είναι ενσωματωμένο σε προϊόντα και εμπορεύματα. Ευχαριστούμε πολύ εκ μέρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπή, ο διευθυντή τη γενική διεύθυνση Κλίματος η κυρία Πετέλσκης. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ε, να ευχαριστήσω τα μέλη του Κοινοβουλίου για αυτό τον επικοδομητικότατο διάλογο που έχουμε σήμερα. Είναι πράγματι πολύ σημαντικό να προχωρήσουμε γρήγορα στην έγκριση αυτής της τόσο σημαντικής πρότασης εν ώψη των ε, διορθωμένων μηνυμάτων που θέλουμε να αποστείλουμε στην αγορά. Για κάποια από τα θέματα που επανήλθαν πολλές φορές στη σημερινή συζήτηση. Πρώτα απ' όλα για την ανταγωνιστικότητα και τη διαρροή του άνθρακα. Νομίζω σε κάθε παρέμβαση θα ακούσαμε αυτά. Θα ήθελα να πω πρώτα-πρώτα ότι οι τομείς που ε, κινδυνεύουν με τη διαρροή του άνθρακα έχουν προστατευθεί από την ε, προσφορά αδειών και αυτό αναγνωρίζεται με τα... Φαίνεται και από τα αποδεκτικά στοιχεία που έχουμε. Το επίπεδο προστασίας είναι εγγυημένο στο τέλος της δεκαετίας. Είναι λοιπόν ε, σημαντικό αυτό για να τοποθετηθούμε στη συζήτηση. Επίσης για την περίοδο μετά το 2020 η δωρεάν ε, απονομή έχει επίσης ε, γίνει έχει πολιτική εγγύηση ως μέρος του πλαισίου 2020 στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να τονίσω ότι είμαστε δεσμευόμαστε μάλλον αυτό να μεταφραστεί και σε νομοθέτημα. Μια νομοθετική πρόταση που να ασχολείται με την, που να καλύπτει την ελεύθερη απονομή και άλλα ζητήματα του ETS μέχρι το 2030 θα είναι έτοιμη πολύ γρήγορα και όλη η σχετική ε, μελέτη θα γίνει συμπεριλαμβανομένων μελετών αντικτύπου. Ξέρω ότι στο σώμα αυτό μεγάλη σημασία δίδεται και στην υψηλής ποιότητας, στις υψηλές ποιότητας μελέτες αντικτύπου. Μετά την έγκριση του ε, αποθεματικού αυτού θα φροντίσουμε να υποβάλουμε πρόταση για την αναθεώρηση του ETS. Αυτή είναι η πρώτη μου παρατήρηση για την ανταγωνιστικότητα και τη διαρροή του άνθρακα. Ως προς τις παραμέτρους, έχω ακούσει πολλές παρεμβάσεις που, συμπεριλάμβαναν, που συμπεριλάμβαναν το στοιχείο αυτό. Να πω τα εξής διαφορετικοί ε, εμπειρογνώμονε δίνουν διαφορετικέ απαντήσει. Αυτό έχουμε ακούσει και στη συζήτηση ω σήμερα. Για το όριο και για το κατά πόσον πρέπει να περνάει κανεί ή να βγαίνει από το αποθεματικό. Κάποιοι θα πούνε μικρότερο ή χαμηλότερο από όσα προβλέπει τώρα η πρόταση τη Επιτροπή. Όμως υπάρχει και η άποψη ότι το φάσμα ορίων που προτείνεται είναι λογικό. Το ακούσαμε και στο εργαστήριο του Κοινοβουλίου, ένα εργαστήριο ειδικών που οργανώθηκε νωρίτερα και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή οργάνωσε επίση ένα εργαστήριο με τη συμμετοχή πραγματομένων τον Ιούνιο. Το αποτέλεσμα τη συζήτηση ήταν λίγο πολύ αυτό. Το αποθεματικό και οι κανόνε τροφοδοσία του αποθεματικού, όπω ε, παρουσιάζονται στην πρόταση τη Επιτροπή, έχουν ε, συνταχθεί και υποβληθεί με μετριοπαθή τρόπο. Μικρά ποσά, μικροί όγκοι θα ε, περιλαμβάνονται αρχικά και για ένα συγκεκριμένο αριθμό ετών. Πριν τα 833 εκατομμύρια ευρώ ως όριο ε, ξεπεραστούν. Πρέπει να ξαναδούμε τη ρήτρα αναθεώρησης ε, που αναφέρθηκε και σήμερα. Η σημερινή ρήτρα αναθεώρησης είναι πενταετής μετά τη θέση σε ισχύ. Θεωρούμε ότι είναι η κατάλληλη στιγμή ώστε να προλάβουμε να δούμε πώς λειτουργεί στην πραγματικότητα το σύστημα και αφού μάθουμε όσα χρειάζεται, προσαρμόζουμε τις παραμέτρους. Αυτή ήταν η προσέγγιση που είχαμε. Πρέπει να, να φροντίσουμε λοιπόν να σταθμίσουμε και να συντάξουμε σωστά τις παραμέτρους και μετά από λίγο καιρό να γίνει αναθεώρηση ε, ε, για την προσαρμογή των παραμέτρων αν χρειάζεται. Η δεύτερη παρατηρήση μετά αυτή και η τρίτη μου είναι για την μετακίνηση της ημερομηνία και τη συμπερίληψη των δικαιωμάτων backload στο MSR. Έχουμε εκφράσει τη θέση μας πολλές φορές και στο Κοινοβούλιο και το έχει πει και ο Επιτροπός μας, ο κύριος Αρίας ήταν σαφής νομίζω. Εάν υπάρξει συμφωνία μεταξύ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου και μετακινηθεί μερομηνία σε νωρίτερο στάδιο, σε πρώτερο στάδιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θα εμποδίσει μια τέτοια πρόταση. Και όπως άκουσα στη συζήτηση νωρίτερα σήμερα, κάποιοι θεωρούν ότι υπάρχουν περισσότερα ωφέλη. Για το αποθεματικό. Αλλά αναφέρθηκε στη συζήτηση ότι θα υπάρξει και μεγαλύτερη σταθερότητα τα τιμών και ότι θα έχουν, αυξηθούν έτσι επενδύσεις στις ε, τεχνολογίες που είναι χαμηλές η κατανάλωση, η κατανάλωση άνθρακα είναι χαμηλή. And I Θα σταματήσω εδώ, Πρόεδρε, και θέλω απλώ να τονίσω και πάλι ότι καλό είναι η πρόταση αυτή να εγκριθεί σύντομα. Mr. Rapporteur, Antonio Tajani. Ευχαριστούμε, συγγητή, ο κύριο Ταγιάννη. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Όπως σας είπα, τη Δευτέρα θα σας παρουσιάσω τη συμβαστική μου πρόταση. Άκουσα πολλά, άλλοι συμφωνούν, άλλοι δεν συμφωνούμε, αλλά τέλος πάντων εγώ συμφωνώ με τα περισσότερα από όσα ακούστηκαν από την Επιτροπή και έχουμε και κάποιες τροπολογίες υποβληθήσεις από τον Ιβο Μπέλετ αυτό σημαίνει ότι μπορούμε ήδη να τα βρούμε με τον ε, εισηγητή της ΕΝΒΗ σε μια πρώτη συμφωνία. Είναι θετικό ότι έχουμε τέτοιες τροπολογίες που υπογράφονται από τον εισηγητή της ΕΝΒΗ. Μένουμε πάντως στο πόσο σημαντικό είναι να φροντίσουμε τον βιομηχανικό ιστό της Ένωσης. Γιατί πολλές φορές είναι εύκολο να αλλάξει κανείς κάποια δημιουργικά στοιχεία ή να φέρει κάτι πιο πιο νωρί πιο αργά, αλλά κατόπιν καταλαβαίνει κανείς ότι από τέτοιε αποφάσεις εξαρτάται η επιβίωση σημαντικών επιχειρήσεων. Και από την εφαρμογή αυτών των κανόνων εξαρτάται η δουλειά χιλιάδων ανθρώπων. Και θα πρέπει να αποφύγουμε ότι στο βωμό του καλύτερου να θυσιάζουμε το καλό. Πολλά από αυτά που άκουσα ε, με βρίσκω σύμφωνο, αλλά, αλλά δεν βοηθούν αναγκαστικά την απασχόληση της επιχειρήσης. Κάνουμε ό,τι μπορούμε, τόσο ώστε να έχουμε όσο γίνεται πιο ευρύ ε, σημαίνηση, να φτάσουμε σε συμβασμούς, όπως είπαμε στην αρχή, και οι σκιώδεις δεν έχουν κάποια αμετακίνητη θέση, κάνουμε ό,τι μπορούμε για να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε συμφωνία. Και να μην αλλάζει, μην αλλοιώνεται η ουσία της πρότασής μου η οποία φυσικά και επιδέχεται βελτιώσει. και για την αναθεώρηση δεν συμφωνώ με τη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η πενταετία ίσως είναι πολύ αντί να κάνουμε κάτι πιο νωρίς αυτή την αναθεώρηση, την επαλήθευση τέλος πάντων τη δοκιμή για την νέα πρόταση και πάντως να προσπαθήσουμε να βρούμε κάτι το οποίο να είναι αποτελεσματικό για τη μείωση των εκπομπών ή για να βοηθήσουμε την παραγωγικότητα και να αποφύγουμε αυτό που είναι διπλός κίνδυνος, δηλαδή με την κατάσταση των επιχείρησεων. Αν θέλουμε να πετύχουμε τους στόχους, και αν δεν μπορούν, τότε θα πάνε εκεί που μπορούν να τους πετύχουν. Και φυσικά τότε θα έχουμε πολλές θέσεις εργασίας. Αυτό δεν πρόκειται να βοηθήσει την βιομηχανία και επίσης πρόκειται και το περιβάλλον να πληγεί. Πάει μια εταιρεία ας πούμε στην Κίνα, καθίσταται Αυτό θα σήμαινε ότι εκεί παράγει με στόχους που είναι πολύ λιγότερο φιλόδοξοι. Ε, και σε ένα περιβάλλον, σε ένα καθεστώς που είναι πολύ λιγότερο αυστηρό. Αυτό να το μην το ξεχνούμε. Τέτοια πρέπει να να κρατήσουμε τις ισορροπίες και η Ήτρε να έχει μια θέση δυναμική γιατί από εδώ ξεκινάει αυτή η υπόθεση. Επομένως, αυτό σημαίνει ότι δεν είναι το οριστικό κείμενο, είναι το κείμενο το οποίο θα πρέπει να δώσει κάποιες κατευθύνσεις δηλαδή το ειδικό βάρος της βιομηχανίας στο γενικότερο πλαίσιο της στρατηγικής. Και κατόπιν έχουμε το οριστικό κείμενο, το τελικό κείμενο το οποίο θα εγκριθεί από την Επιτροπή Περιβάλλοντος και που θα πρέπει να λάβει υπόψη όλες τις απόψεις, όλες τις πλευρές για τη βιομηχανία και το περιβάλλον. Άρα, ως Επιτροπή Βιομηχανίας θα πρέπει να μην σκεφτόμαστε 100% την ε, βιομηχανία ε, θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας την βιομηχανία και κατόπιν η ένβη ελπίζω να λάβει υπόψη τις προτάσεις μας και να διατυπώσει πρόταση ούτω ώστε να μπορέσουμε να παντρέψουμε τα διάφορα συμφέροντα τα, τα μεταξύ δηλαδή της πολιτικής για την αλληλεγγύη του κλίματος και τα της επανεκβιομηχάνησης. Σας ευχαριστώ για προτάσεις και για ιδέες. Με προσοχή τα άκουσα. Όλα αυτά θα τα ζυγίσουμε υπό και τις τροπολογίες σας. Το ότι έχουμε τόσες προτάσεις αυτό σημαίνει ότι ενδιαφέρεστε. Γιατί είναι πολύ σημαντικό το θέμα για όλους. Θα προσπαθήσω να εισηγηθώ κάποιες προτάσεις που θα συγκεράσουν τις επιμέρους διαφορετικές θέσεις. Θα συζητήσουμε και με τον Μπέλετ. Ε, μας τα είπε και ελπίζουμε ότι αυτό θα διαμορφώσει το τελικό κείμενο, το οποίο θα το συνδιαμορφώσει και η Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα λοιπόν θα περιμένουμε... Αναμένουμε οι συναδελφοί μας από την Επιτροπή Περιβάλλοντος να λάβουν την υποδότησή μας πολύ σοβαρά θα εγκρίνουμε το σχέδιο γραμματότησης στις 22 Ιανουαρίου, 22 Ιανουαρίου 2015. Η ψηφοφορία στην Επιτροπή Περιβάλλοντος θα γίνει στις 24 Φεβρουαρίου του 2015. Ένα μήνα λοιπόν αργότερα περίπου. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ τον εισηγητή, τους Κιώδης και όλους τους συναδέλφους της πολύ σπουδαίας αυτής της συζήτησης. Και τώρα να περάσουμε στο τελευταίο σημείο στην ημερήσια διάταξη, η οποία ήταν βαρυφορτωμένη αυτή τη φορά. Πάμε λοιπόν στο σημείο υπαριθμό 12. μετά το σημείο 11 αλλά και μετά το σημείο 13. 2015. Σχεδιασμός για το Διεθνή Χάρτη Ενέργειας 2015 παρουσίαση από τον Γενικό Γραμματέα του Χάρτη Ενέργειας του δόκτωρα, τον δόκτωρα Ούρμπαν Ρουσνάκ. Επιτρέψτε μου να τον καλωσορίσω. Σας ευχαριστούμε που ήλθατε. Μας ενδιαφέρει πολύ τι γίνεται και ποιες είναι οι εξελίξεις σε ό,τι αφορά το χάρτη ενέργειας σε παγκόσμιο επίπεδο. Η πολιτική κρίση στην Ουκρανία κατέδειξε πόσο σημαντικό είναι το ζήτημα αυτό, το θέμα της ασφάλειας της ενεργειακής προμήθειας και παροχής. Γνωρίζουμε την ανακοίνηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ενέργεια που δημοσιεύτηκε το Μάιο και τη συμφωνία του Συμβουλίου για τις ε, πολιτικές για τις ενέργεια που δηλώνει ότι η ενεργειακή αποδοτικότητα, οι ανανεώσιμες και η ενεργειακή ασφάλεια, η επάρκεια θα πρέπει να συμπεριληφθούν σε όλες μας τις σχέσεις με... που έχουν να κάνουν με την ενεργειακή πολιτική. Τελευταίο σημείο στην ε, δήλωση αυτή την προκαταρτική. Θα ήθελα να πω ότι η συνεχιζόμενη εργασία της Ήτρε για την ε, έκθεση ίδιας πρωτοβουλίας με εισηγητή τον κύριο Σαοντάργας για την στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ενέργεια είναι πολύ σημαντική. Διοργανώθηκε λοιπόν και σχετική ακρόαση σε ό,τι αφορά θέματα ενεργειακής ασφάλειας. Έγινε χθε και μία ανταλλαγή απόψεων για την έκθεση ίδιας πρωτοβουλίας. Κύριε Ρούσνεκ, αν θα θέλετε να πάρετε το λόγο για να μα παρουσιάσετε και τη δική σας τοποθέτηση. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μέλη του Κοινοβουλίου, είναι τιμή μου να απευθυνόμαι στην Επιτροπή Ενέργειας και Έρευνας και τεχνολογία σήμερα στο Κοινοβούλιο. Εδώ ήθελα να σας μιλήσω για, την, ε, για τον χάρτη της ενέργειας και το τη διαρκή διαδικασία εξυγχρονισμού του. Να σας ευαισθητοποιήσω στο θέμα αυτό. Πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Ένωση άρχισε να συζητά για το πώς θα πρέπει να προχωρήσει σε μια ενεργειακή ένωση. Να σημειώσω ευθύ εξ αρχής ότι η διαδικασία του χάρτη ενέργειας και η Ενεργειακή Ένωση βρίσκουν ε, το έναυσμά τους στις αρχικές προτάσεις του Ολλανδού Πρωθυπουργού ε, Λούμπεκ από το 1990 για ενεργειακές κοινότητες. Και νομίζω ότι είναι σημαντικό, σημαντικό να ξέρετε πώς έχει ξεκινήσει αυτή η διαδικασία για το Διεθνή Χάρτη Ενέργειας με τις δηλώσεις σχετικά με το χάρτη αυτό. Πριν μιλήσω για τον εξυγχρονισμό, την επικαιροποίηση του χάρτη, να τονίσω δύο σημαντικά ζητήματα. Αναφερόμαστε στον χάρτη ενέργειας για δύο λόγους. Πρώτα απ' όλα, για μια πολιτική δήλωση του 1991 που ονομάζεται Ευρωπαϊκή, ε, Ευρωπαϊκός χάρτης ενέργειας, μια πολιτική δήλωση που εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση των 12 τότε. Και με χώρες ε, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, της τότε Ανατολικής Ευρώπης και άλλες χώρες της Ευρασίας, οι Πολιτείε, Πολιτείες λόγω χάρη. Ε, οι υπόλοιποι ε, εξαιρέθηκαν από την δήλωση αυτή. Έπειτα, στη Λισαβόνα ε, εγκρίθηκε η επόμενη φάση του χάρτη. Κάθε ε, κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν ε, συμβαλόμενο μέρος στην σύμβαση αυτή. Το 1991 όταν εγκρίθηκε ο Διεθνής Χάρτης για την Ενέργεια ξεκίνησε η διαδικασία. Και το 1994 υπογράφηκε όπως είπα η σχετική συνθήκη. Τέθηκε σε ισχύ το 1998 και έχει κυρωθεί πλέον από 52 χώρες η συνθήκη αυτή. Τρεις χώρες είναι αυτή τη στιγμή στην διαδικασία ε, ε, κύρωσης. Το Μαυροβούνιο, η Γεωργία και το Πακιστάν. Η Ρωσική Ομοσπονδία, η Λευκορωσία, η Ισλανδία, η Νορβηγία και η Αυστραλία δεν έχουν κυρώσει τη συνθήκη ακόμη. Ο ενεργειακός χάρτης λοιπόν ελέγχεται από τη διάσκεψη του χάρτη που ασχολείται με όλους τους ενεργειακούς χάρτες. Βασικός ρόλος του σώματος είναι να ε, παρακολουθεί την εφαρμογή και τις δεσμευτικές ε, αρχές των ενιών και των αρχών του χάρτη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι συμβαλλόμενο μέρος και εφόσον το αποφασίσει η διάσκεψη και άλλα κράτη εκτό συνθήκη μπορούν να προσκληθούν ω παρατηρητέ. Τι ε, προσφέρει αυτή η συνθήκη. Η συνθήκη έχει περισσότερα από 50 μέλη όπω ανέφερα και βασίζεται σε δύο αρχέ. Την εθνική κυριαρχία για του ενεργειακού πόρου, που είναι πολύ σημαντική για τις ε, ενεργειακά πλούσιε χώρε και μετά η προστασία τη ενέργεια βάσει τη μη διακριτικής μεταχείρισης. Σημαντική για τι χώρε που επενδύουν στις ενεργειακά πλούσιες χώρες. Ως προς το εμπόριο, ο χάρτης βασίζεται στους κανόνες του ΠΟΕ, που όπως ξέρετε δεν έχει καμία συμφωνία για την ενέργεια στο επίπεδο του ΠΟΕ. Συμπληρώνει λοιπόν αυτό το κενό των κανόνων του ΠΟΕ για το εμπόριο ενέργειας ε, ο χάρτης. Η συνθήκη προβλέπει και ένα μηχανισμό επίλυσης διαφορών ISDS ή μεταξύ κρατών μέρος του, της ε, συνθήκης ασχολείται με την ενεργειακή αποδοτικότητα που περιγράφεται στο πρωτόκολλο για την ενεργειακή αποδοτικότητα καθώς και παρακολουθεί τις εξελίξεις στην αγωγή ενέργειας. Τι έχουμε εκδώσει ως τώρα, κάποια ήπια εργαλεία για τους επενδυτές και τα συμβαλόμενα μέρη με μια σύγχρονη ε, συμφωνία για την ταχεία οικοδόμηση διασυνοριακών υποδομών ή για το μηχανισμό έγκαιρης προειδοποίησης. Κάτι που επιτρέπει στα συμβαλόμενα μέρη της Υπηρεογειακού Χάρτη του 1991 να αντιδράσουν εφόσον χρειαστεί. Για τον εξυγχρονισμό τώρα της, ε, του χάρτη, όταν ξεκίνησε το 2012 ε, διάσκεψη. Η πρώτη της ε, σύνοδος οργανώθηκε στη Βαρσοβία. Και τότε συζητήσαμε την εντολή για την γεωγραφική ε, εξάπλωση του χάρτη με τη συνθήκη να συμπεριλαμβάνει πλέον την πολιτική δήλωση για τον ενεργειακό χάρτη του 1991, το 2014. Ήδη άρχισαν να συζητώνται οι παράμετροι του νέου χάρτη και το 2014. Το 2013 μάλλον συζητήθηκαν ξανά οι τέσσερις βασικές αρχές του χάρτη και το 2014 όλα τα συμβαλόμενα μέρη συμμετείχαν στις συνόδους μαζί με νέα μέλη που προσκλήθηκαν να συμμετέχουν στη διαδικασία του χάρτη. Ποιο, ποια θα μπορούσαν να είναι τα μέλη της διαδικασίας του ενεργειακού χάρτη εφόσον υπάρξει διεύρυνση. Από την περιοχή του Ειρηνικού και του της Ασίας, η Ινδονησία υπέγραψε το χάρτη το 2009, οι χώρες της ΑΖΕΑΝ, της Νότιας Ασίας, ε, και της συνεργασίας της Νότιας Ασίας. Επίσης, η Κίνα τη τη για τον ενεργειακό χάρτη για να ενισχύσει τις σχέσεις της ε, με τον χάρτη και εκεί έχουμε δει να επιτυγχάνεται πρόοδος στις σχέσεις μας. Με τη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική, την νότια γειτονιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνεργαζόμαστε στενά με τις χώρες της Αφρικής και με την Μέση Ανατολή για να κυρώσουν τον χάρτη και βλέπουμε αυξανόμενο ενδιαφέρον και από λατινοαμερικανικές χώρες. Ιδίως αυτές που στις οικονομικές τους πολιτικές προωθούν την ελεύθερη αγορά. Μεξικό, Κολομβία, Χιλή ή Περού. Στην Αφρική βλέπουμε επίσης αυξανόμενο ενδιαφέρον, νοτίως της Σαχάρας, από τη Μαυριτανία ή χώρες που έχουν ήδη εκφράσει ενδιαφέρον όπως ο Νίγηρας, η Νιγηρία, η Μοζαμβίκη, η Τανζανία και η Αγγόλα. Βλέπετε ότι αυτές οι χώρες είτε ήδη είναι παλιή παραγωγή ενέργειας είτε προορισμοί. Να προσθέσω μερικές ε, σύντομες ε, φωτογραφίες, ε, συνοπτικές παρουσιάσεις για το για τις αρχές της ε, του χάρτη. Ήθελε να βελτιώσει την ενεργειακή επάρκεια ο χάρτης αρχικά όταν ε, εγκρίθηκε, κυρίως να σταθεροποιήσει τις σχέσεις ε, Βρυξελών-Μόσχας. Σιγά σιγά όμως αρχίσαμε να πηγαίνουμε προς τον Νότο. Και υπάρχουν λόγοι γι' αυτό. Νομίζουμε η απάντηση για την ενεργειακή επάρκεια στη διαδικασία του χάρτη είναι να δημιουργηθεί ένα περιβάλλον κατάλληλο για τις επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες. Είναι σημαντικό αυτό και για τις κυβερνήσεις και για τους επενδυτές, για να υπάρχει σωστή ισορροπία μεταξύ υποχρεώσεων και μακροπρόθεσμων δεσμεύσεων στις ενεργειακές επενδύσεις. Ε, χρειάζεται μια αποτελεσματικότερη ενεργειακή αγορά, διότι η περιφερειακή ενεργειακή συνεργασία είναι κλειδί για την επιτυχία. Δεν υπάρχει λύση για καμιά χώρα μεμονωμένα στον κόσμο και βλέπουμε ότι η παγκοσμιοποίηση της αγοράς ενέργειας προχωρά πολύ γρήγορα. Δεν υπάρχει καμία χώρα που μόνη της μπορεί να λύσει τα ενεργειακά της προβλήματα. Χρειάζεται λοιπόν ε, περιφερειακή και βασισμένη στην αγορά συνεργασία. Για την ενεργειακή αποδοτικότητα επίσης είναι πολύ σημαντικός ο χάρτης, διότι το κόστος της ενέργειας είναι υψηλό ε, υπάρχουν κλιματικές αλλαγές και άλλες προκλήσεις ε, που ε, θέτουν ένα την ενεργειακή επάρκεια. Ο καλύτερος λοιπόν τρόπος είναι η αποδοτικότητα. Έτσι αντιμετωπίζονται οι προκλήσεις αυτές. Το ίδιο και με την ασφάλεια και την ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών προβλημάτων. Συγγνώμη. Τα είπατε και στην Επιτροπή σας πριν την παρουσίασή μου. Είναι πολύ σημαντικό στο πλαίσιο της συνθήκης για τον χάρτη της ενέργειας, αλλά και στα πλαίσια των μηχανισμών επίλυσης διαφορών για διατησίες μεταξύ κρατών, σε διαφορές μεταξύ κρατών ε, και μηχανισμούς διατησίας μεσολάβηση σε περίπτωση που εμπλέκονται και επενδυτές ή την, ε, τον συμβιβασμό όσων μπορεί να ε, είναι διάδικοι σε περιπτώσεις που έχουμε αγωγούς που περνούν από περισσότερα του ενός κράτη. Τι απαιτείται τώρα. Με την υποδοχή της κυβέρνησης της Ολλανδίας ελπίζουμε ότι θα διοργανωθεί ε, και θα προκύψει μια διεθνής δήλωση του χάρτη που αν όλα πάνε καλά θα υπογραφτεί στη Χάγη τον Μάιο του 2015. Έχετε δει το σχέδιο κειμένου, αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων μεταξύ των συμβαλωμένων μερών και όσων συμμετέχουν για πρώτη φορά. Αναζητούμε την πολιτική στήριξη από τα κράτη-μέλη και την Ευρωπαϊκή Ένωση γενικότερα. Είναι καθοριστική σημασία σε αυτό, γιατί πρέπει όλα αυτά να γίνουν πραγματικότητα. Η βασική αρχή και ο βασικός λόγος που προσπαθούμε να κάνουμε τις αρχές και τους κανόνες της, ε, του ενεργειακού χάρτη διαθέσιμο σε διεθνέ επίπεδο είναι ότι εδώ υπάρχει ένα τεράστιο περιθώριο ευκαιριών. Οι νέε ενεργειακές αγορές να δεχτούν τις ευρωπαϊκού χαρακτήρα αρχές μας. Εάν αποτύχουμε και δεν έχουμε μεγαλύτερη στήριξη σε διεθνές επίπεδο, η ενεργειακή συνεργασία με αρχές που να συμπεριλαμβάνονται στις βασικές νομοθετικές δομές της Ένωσης και των κρατών μελών, θα πρέπει η Ένωση και τα κράτη της να προσαρμοστούν σε νέους κανόνες που θα έχουν προκύψει από τα φυτόρια παραγωγής ενέργειας σε διαφορετικά μέρη του κόσμου. Θα σταματήσω εδώ, Πρόεδρε, και είμαστε διαθέσιμοι για ερωτήσεις. Uh, thank you, Σας ευχαριστώ, Δόκτωρα, για την παρουσίασή σας. Συνάδελφοι. Αν θα θέλετε να κάνετε σχόλια. Ο συνάδελφος Ρούμπιχ. Να ευχαριστήσω γιατί ο χάρτη ενέργειας παίζει καθοριστικό ρόλο και θα παίξει καθοριστικό ρόλο για τη συνεργασία μας στο μέλλον. Και γι' αυτό πιστεύω ότι από πλευρά Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μας ενδιαφέρει ιδιαίτερω να παρακολουθήσουμε τις εξελίξεις και να δούμε που υπάρχει περιθώριο βελτίωσης. Ιδιαίτερα σε καιρούς όπως η σημερινή, όπου η ενέργεια είναι στο επίκεντρο της πολιτικής προσοχής οι συγκρούσεις θα πρέπει να προλαμβάνονται εξ αρχής και να υπάρχει καλύτερη συνεργασία. Πώς μπορεί λοιπόν να γίνει αντιληπτή η πολιτική κατάσταση, υπάρχουν από πλευρά σας συγκεκριμένες επιθυμίες. Ο συνάδελφος Κέλλη. Σας ευχαριστώ. Προφανώς η τιμέ της ενέργειας θα είναι και σημαντικές, σημασία σημασίας για την Ευρώπη στο μέλλον, για να επαναβιομηχανοποιηθεί η Ευρώπη. Και γι' αυτό λοιπόν θα είναι σημαντικός ο χάρτης ενέργειας. Σε ό,τι αφορά την επίθεση της Ρωσίας στα σύνορά μας προς Ανατολάς, πώς επηρεάζει αυτό το χάρτη της ενέργειας, τι μπορεί να γίνει λοιπόν για να επιληθούν τα ζητήματα που ε, επηρεάζουν ιδιαίτερα την ασφάλεια εφοδιασμού και φυσικά και το κόστος της παροχής. Σας ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Να σας ζητήσω, κύριε Γενικά Γραμματέα, να απαντήσετε στις, ε, συγγνώμη, και στις δικές μου ερωτήσεις. Καταρχάς, σε ό,τι αφορά την πλήρη συμμόρφωση όλων μας των κανονισμών στην Ευρωπαϊκή Ένωση εσωτερική αγοράς. Το πακέτο της ενεργειακής, ε, του ενεργειακή χάρτη. Ελπίζω λοιπόν όλα αυτά να συνάδουν 100%. Θα ήθελα όμως και τη δική σας άποψη ως επαγγελματία. Και κατά δεύτερον, η δυνατότητα υποστήριξης των χωρών ενεργειακής κοινότητας. Ε, 8 χωρών, Σαββατικά Βαλκάνια, Ουκρανίας, Μολδαβίας, Γεωργίας, για να αξιοποιηθεί η συνθήκη του ενεργειακού χάρτη, γιατί συχνά βρίσκονται σε δύσκολη θέση σε ό,τι αφορά τους εξωτερικούς παρόχους και προμηθευτές. Προσπαθούμε λοιπόν να τους βοηθήσουμε. Πώς μπορούμε λοιπόν να το πράξουμε αυτό με βάση τη συνθήκη. Ποια είναι η άποψή σας. Δεν έχουμε άλλες ερωτήσεις, λέει ο κ. να απαντήσω τώρα. Εμείς συνεργαζόμαστε με την υπηρεσία εξωτερικής δράσης και με την Επιτροπή. Πάρα πολύ εύστοχη ερώτηση γιατί όπως σας είπα τώρα έχουμε τη διαδικασία της διεύρυνσης του ενεργειακού χάρτη. Έχουμε περιορισμένες, περιορισμένους ανθρώπινους πόρους στην γραμματεία είμαστε περίπου 30 και ελπίζουμε ότι στη συνέχεια με τις επαφές με τα θεσμικά όργανα θα υποστηριχτούμε. Ε, σε επίπεδο διπλωματίας ευρωπαϊκής και ότι ο χάρτης πρόκειται να προωθηθεί μέσω των διπλωματικών διάβλων της υπηρεσίας εξωτερικής δράσης. Επίσης άλλη πλατφόρμα, άλλο, άλλο φόρουμ που να κινηθούμε είναι το, η G20. Τώρα όσον αφορά την βιομηχάνηση, μηχάνηση της ε, Ευρώπης και τις σχέσεις με την Ανατολή και την Ρωσία, αυτό έχει σχέση και με τις τελευταίες ερωτήσεις του Προέδρου και θα ήθελα να σας ε, διευκρινίσω ότι η Ρωσία προσωρινά μεταξύ 1994 και 2009 εφήρμοζε τη συνθήκη το 2009 σταμάτησε, απεσύρθη. Και ο λόγος που αυτό έγινε είναι, είναι πολύ. Όμως υπήρξαν αποφάσεις 2003-2004 από κυβερνήσεις όσον αφορά την απαλωτρίωση στοιχείων περιουσιακών της Γιούκος κατόπιν ε, παραβιάσεων της συνθήκης. Είχαμε επιδιαιτησία, κράτησαν 10 χρόνια και παραπάνω, τελειώσαν το καλοκαίρι, οπότε και η Ρωσία καταδικάστηκε να πληρώσει αποζημίωση στους επενδυτές της Γιούκος 50 δις δολάρια. Βαρύτερη χειρματική ποινή ποτέ έχει επιβληθεί από, ε, από το χάρτη από οποιαδήποτε άλλη συνάφη ε, συνθήκη. Δεν έγινε ποτέ αυτό γιατί ζήτησε να ανασταλεί η ισχύ της απόφασης και η εκτέλεσή της ε, η Ρωσία. Αλλά πολύ σημαντικό στοιχείο αυτό για το μέλλον γιατί αποτελεί στοιχείο υλοποίησης του χάρτη. Και οι επενδυτέ θα ζητήσουν να παγώσουν τα στοιχεία του ενεργητικού ε, της Ρωσίας ε, των ρωσικών ε, εταιριών. Υπάρχει αστάθεια επομένως σε αυτό το σημείο. Τώρα όσον αφορά την ε, ασφάλεια της διμετακόμισης με, από τον αγωγό που περνάει από την Ουκρανία, το σημαντικό στοιχείο του χάρτη ενέργειας είναι το ότι δεν υπάρχει εδώ κάποιο πρόβλημα, κάποια αμφιβολία, αλλά από το 2006-2007 τον έχουμε τον χάρτη σαν ένα εργαλείο στη διάθεσή μας και εξαρτάται από τα συμβαλόμενα μέρη, το αν θέλουν να το χρησιμοποιήσουν αυτό ε, το, το χάρτη, το, το εργαλείο. Δεν είχε χρησιμοποιηθεί με το 2014. Οι χώρες προσπάθησαν να κάνουν κάποιο είδου συμφωνία. Έξω νομική τέλος πάντων. Για να μην χρησιμοποιήσουν αυτό το εργαλείο που έχουν στη διάθεσή τους και πιστεύω ότι αυτό όσο θα χρησιμοποιηθεί το 2009 τότε που είχαμε επίλυση άλλων διαφόρων σε πολιτικό επίπεδο και η κατάσταση αν είχε γίνει αυτό θα ήταν σήμερα ασφαλέστερη πιο προβλέψιμη γιατί οι ρίζες της κρίσης βρίσκονται πίσω στο 2009 τότε που ξεκίνησε η, κρίση του φυσικού Τώρα όσον αφορά την ε, συμμόρφωση με την ε, ε, με τη συνθήκη όπως ξέρετε όταν είναι πολύ νομική ο καθένας και του άποψη και όσον αφορά τη Ρωσία εκεί ο χάρτης σταμάτησε να ισχύει το 2009, δεν, δεν την προσέβαλαν, δεν προσέβαλαν το χαρτί επισήμω. Άρα ε, δεν ξέρουμε ακόμα τι θα αποφασίσει κάποιο ανεξάρτητο δικαστήριο. Δεν ξέρουμε εάν η, ο χάρτης έρχεται σε σύγκρουση με, το, με τη δέσμη ενεργειακών μέτρων όπως έχουν πει κάποιοι Ρώσοι. Πάντως, σύμφωνα με δικές μας αναλύσεις, πώς να το πω. Δεν ξέρουμε, επί ξηρού ακμής βρισκόμαστε για το τι θα γίνει με την ε, εφαρμογή, τι θα γίνει, ε, αν, θα υπάρξει ή όχι παραβίαση του χάρτη. Αυτό θα προκύψει από την ε, διαδικασία. Άρα κρεμεί το θέμα. Τώρα όσον αφορά το να εξασφαλίσουμε την ενεργειακή ασφάλεια για τις ε, χώρες της όμορες τη συνθήκη συνθήκη να προσχωρήσει στη Σερβία και το Μαυροβούνιο. Είναι πολύ σημαντικό στοιχείο για την ενεργειακή ασφάλεια πάντως το να έχουμε σταθερότητα, να έχουμε επενδυτικό καλό κλίμα δεν σχετίζεται άμεσα με την ε, ενδιακή ασφάλεια, αλλά θα πρέπει να ισχύουν οι κανόνες του παιχνιδιού. Οπότε και έτσι όλες οι χώρες που συμμετέχουν, όλα τα συμβαλώμενα μέρη, εάν κάνουν αυτό που πρέπει, τότε το σύστημα αποδίδει. Εάν κάποια χώρα δεν θέλει να εφαρμόσει και να συμμορφωθεί, τότε μπορούμε να πιέσουμε κι εμείς Αλλά αυτό δεν γίνεται άμεσα. Άρα σε απάντηση ότι σας πρόεδρε, η προσχώρηση της ε, Σερβίας στον χάρτη, όπως και το Μοντενέγκρο, θα συμπληρώσει το μοσαϊκό. Δηλαδή ότι όλες οι χώρες των Βαλκανίων θα είναι υπό τις ίδιες συνθήκες στον χάρτη. Έχουμε και την Γεωργία από το 2015 πρόκειται να κυρώσει τη συνθήκη. Και έτσι θα επικραθεί το κεκτημένο. Ό,τι χρειάζεται το έχουμε. Αλλά χρειάζεται πιο επιδέξια χρήση αυτών των μέσων και εργαλείων από την διοίκηση αλλά και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ κύριε Γενική Γραμματέα, λέει ο Ευχαριστήσουμε. Και ευτυχώ, επειδή έλειπαν ε, πολλά μέλη τη Επιτροπή μα, είχα την ευκαιρία να θέσω και εγώ κάποιε ερωτήσει. Ήταν εξαιρετικό αυτό, γιατί συχνά τον έρχεται ο χρόνο. Θα ήθελα κλείνοντα να πω ότι είναι εξαιρετικό το έργο του Γενικού Γραμματέα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προστοσία σας. Κυρίε και κύριοι, θα ήθελα να πω δύο λόγια στη μητρική μου γλώσσα. Οι διερμηνείς μας μας συνόδευσαν επί δύο ημέρες. Θα ήθελα ευγενικά να τους ευχαριστήσω και να ευχαριστήσω τους διερμηνείς της πολωνικής καμπίνας και να τους πω ότι τους άκουγα όλη την ώρα. Το κανάλι παριθμών 18. Δεν ακούω αγγλικά, κάποια φορά μιλάω φυσικά αγγλικά, αλλά πάντα ακούω την καμπίνα παριθμών 18. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή στη συνεδρίαση αυτή. Στις 5 υπολογίζαμε ότι θα κλείναμε τη συνεδρίασή μας και όπως βλέπετε η ώρα είναι 17.00. Παρά το γεγονός ότι αλλάξαμε την ημερήσια διάταξη, τελειώσαμε στην ώρα μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ε, εργασίες μας φέτος. Η επόμενη συνεδρίαση της, ομα... της Επιτροπής μας θα λάβει χώρο την επόμενο έτος. Ευχαριστώ πολύ και τα του χρόνου.